Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Και Όλοι παρακαλώ, αν έχετε την ευγενή καλεσύνη να μπείτε ησύχω για να ξεκινήσουμε και τι εργασίε. Allora, buongiorno a tutti. Eh, Καλημέρα σε όλους. Ξεκινούμε με το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Τα όσα αποφασίστηκαν στους συντονιστές εχθές στις εργασίες της συνεδριασής μας. Οι συντονιστές εχθές αποφάσισαν να εγκρίνουν την πρόταση προφορικής ερώτησης για την αναφορά 901-2008 που παρουσίασε ο David ε, Skinner για την ελευθερία του μη συνεταιρίζεστε. Επίσης συμφώνησαν για την πρόταση ερώτησης για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην έκθεση Auken για τον ε, νομοθεσία των ακτών στην Ισπανία κατόπιν ετήσεων τη αναφορά 159-2010 που παρουσίασαν οι κυρίε Χίλεν και Πράιορ και αποφάσισαν να αναστείλουν την ε, απόφαση και να περιμένουν να ληφθεί απόφαση μετά από τη συζήτηση που θα γίνει σήμερα για τις ε, πολυάριθμες αναφορές που έχουν ως αντικείμενο το ίδιο θέμα, δηλαδή τον ε, νόμο των ακτών της Ισπανίας. Για το σημείο αυτό, το οποίο προβλέπει και μία συζήτηση για πάρα πολλές αναφορές στη σημερινή συνεδρίαση, οι συντονιστές αποφάσισαν να κατατάξουν τις εργασίες ε, κατά σειρά ώστε να δώσουν τη δέουσα προσοχή και να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη συζήτηση. Αποφασίστηκε λοιπόν στους 30 περίπου αναφέροντες ε, που είναι παρόντες ε, να δοθεί ο λόγος στην έναρξη της συζήτησης σε 9 εκπροσώπους από διάφορες ε, περιοχές της Ισπανίας. Με άλλα λόγια, αποφασίσαμε να ομαδοποιήσουμε τις αναφορές ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Επειδή είναι πάρα πολλοί από τους αναφέροντες παρόντες, θα δοθεί ο λόγος για τρία λεπτά στον καθένα και στη συνέχεια μετά από τις παρεμβάσεις και των ε, ε, αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ξεκινήσει η συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής ε, που θα φροντίσουν και αυτοί, σας παρακαλώ, να περιορίσουν τις παρεμβάσεις τους στο ένα λεπτό. Όσον αφορά τώρα το σημείο υπαριθμών 3 στην ημερήσια διάταξη των συντονιστών, αποφασίσαμε να συσταθεί μια ομάδα εργασίας που θα ασχοληθεί με τη δημιουργία ενός πλαισίου για τα θέματα που άπτονται του Jugendamt και τις σχετικές αναφορές. Οι συντονιστές αποφάσισαν να ε, παρουσιάσουν έναν υπεύθυνο από κάθε ομάδα και αποφασίστηκε ότι τα μέλη αυτής της ομάδας εργασίας ε, στη συνέχεια θα είναι και τα μέλη της αντιπροσωπείας η οποία θα μεταβεί στο Βερολίνο στα τέλη Ιουνίου. Για το σημείο αυτό των επισκέψεων θα ήθελα να προσθέσω ότι οι αιτήσει για επισκέψεις και στη Βουλγαρία και στο Βερολίνο έγιναν δεκτές, επομένως αποφασίσαμε να κάνουμε και τις δύο αποστολές στα τέλη Ιουνίου, όπως ε, προτείνει και το Προεδρείο, γιατί τότε είναι η πιο κατάλληλη ευκαιρία και για να μην υπάρχει και αλληλοεπικάλυψη με τις ε, εργασίες του Κοινοβουλίου. Θα γίνει λοιπόν η επίσκεψη στη Βουλγαρία όπως ε, έχει διανεμηθεί και στο πρόγραμμα στις 29 Ιουνίου και ταυτόχρονα θα έχουμε και την επίσκεψη στο Βερολίνο και αυτή βάσει του σχεδίου προγράμματος που σας έχει διανεμηθεί, το οποίο όμως ακόμα πρέπει να οριστικοποιηθεί για κάποιες λεπτομέρειες. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συντονιστές λοιπόν να μας πούνε ποιοι θα συμμετέχουν στις δύο ομάδες και στις ε, δύο αντιπροσωπείες στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης ε, για την ε, πρωτοβολία των πολιτών. Σας έχει δοθεί μία επιστολή την οποία θα αποστείλω στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου για να υπενθυμίσω τη δέσμευση που αναλάβαμε στη διάρκεια της έγκρισης του κανονισμού για την πρωτοβουλία αυτή να δώσουμε δηλαδή την δυνατότητα στην Επιτροπή Αναφορών με μια συγκεκριμένη ε, τροποποίηση στον κανονισμό την αρμοδιότητα για να κάνει την ακρόαση ε, όσων θα παρουσιάσουν τις ε, πρωτοβουλίες των πολιτών για την οργάνωση σεμιναρίου για την εφαρμογή της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, θέμα για το οποίο αποφάσισε να ασχοληθεί η Επιτροπή. Εχθές ε, σας είπα ότι ξεκίνησε και αντίστοιχη διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της αρμόδιας Επιτρόπου Ρέντινγκ μας ε, ενημέρωσε ότι ξεκινά η οργάνωση μιας μεγάλης ε, δημόσιας διαβούλευσης επί του θέματος και όπως προβλέπεται από τον κανονισμό ο οποίος ενεκρίθη θα διοργανωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με την Επιτροπή Αναφορών. Εχθές, στη διάρκεια της συνεδρίασης των συντονιστών, αποφασίσαμε να δεχτούμε την ε, πρόσκληση που διατυπώνεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να επιλέξουμε και τους προσκεκλημένους που θα, ήθελα, θα θέλαμε να συμμετάσχουν. Έχουμε προτείνει επίσης να συμμετέχει και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών γιατί είναι και δική της αρμοδιότητας το θέμα και από εκεί και πέρα να οργανώσουμε το σεμινάριο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μην ε, ε, κάνουμε την ε, ανεξάρτητη πρωτοβουλία που είχαμε αποφασίσει εμείς ως Επιτροπή Αναφορών. Τέλος, ακούσαμε την ανακοίνωση της Αντιπροέδρου Παλιαδέλη εχθές για την αίτηση να απαντήσουμε σε ένα ερωτηματολόγιο που ετοίμασε η Επιτροπή Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών. Η κυρία Παλιαδέλη ετοίμασε και μία απάντηση την οποία μας παρουσίασε και έχει διανεμηθεί και σε όλα τα μέλη για τις ερωτήσεις ε, που έχει θέσει η Επιτροπή Γυναικών. Στη συνέχεια εγκρίναμε και την ημερήσια διάταξη για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας με δύο τροποποίησεις, δύο επιπλέον σημεία προσετέθησαν δύο θέματα που είχε ζητήσει η ομάδα των σοσιαλιστών. Δεν συζητήθηκε κάτι άλλο. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις και δεν θέλει κάποιος το λόγο, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε απευθεία στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης έχουμε ψηφοφορία. Θα ξεκινήσει λοιπόν τώρα η ψηφοφορία. Κολέγα θα ήθελα να κάνω μία σύντομη εισαγωγή. Καταρχήν, θεωρώ... Μισό λεπτό. Να συζητήσουμε, να, να σας αναφέρω και ποιο θέμα θα συζητήσουμε στην ημερήσια διάταξη. Μισό λεπτό, κυρία Όκεν. La, la collega vuole illustrare il... Η κυρία Άουκεν θέλει να παρουσιάσει το έγγραφό τη, έτσι δεν είναι, αυτό δεν θέλετε να κάνετε. Μισό λεπτό, διότι πρώτα έχουμε την γνωμοδότηση Τσίτσεστερ, μετά έχουμε τη δική σας τη γνωμοδότηση και πριν ξεκινήσουμε την πληροφορία, ούτως ή άλλως δίνω το λόγο στους συντάκτες. Μισό λεπτάκι. Sul 13. Σημείο υπαριθμών 13. Γνωμοδότη σχετικά με την κινητικότητα και την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία. Συντάκτη ο κύριο Τσίτσεστερ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τσίτσεστερ αν θέλει να λάβει το λόγο. Yes, thank you, Madam Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο σημεία. Ευχαριστώ καταρχήν του συναδέλφου ε, για τι εισφορές, τι τροπολογίε που έχουν υποβάλει σε αυτή τη γνωμοδότηση. Μεγάλη πλειοψηφία αυτών ε, έχουν γίνει δεκτέ, τι υποστηρίζω μία τροπολογία έχει υποβληθεί δύο φορές τον ίδιο συνάδελφο. <clears throat> Θα δείτε ότι σε ένα σημείο την έχω δεχτεί, αλλά θεωρώ ότι δεν ε, είναι αναγκαίο να δεχτώ την τροπολογία 2, μότι και 14. Εγώ έχω δεχτεί την 2 και προτείνω να απορρίψουμε την 14 γιατί είναι το ίδιο ε, κείμενο. Ευχαριστώ πολύ και τη Γραμματεία για την βοήθειά της. Ευχαριστούμε κύριε Τσίτσεστε. Να ξεκινήσει η ψηφοφορία λοιπόν. Τροπολογία 1, παράγραφος 1, από την ε, κυρία Κίνγκα Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 1, τροπολογία 2, Τιτσιάνο Μότι. Ψηφοφορία κατά τμήματα για τις δύο παραγράφους. Ε, άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν για την πρώτη παράγραφο υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3, παράγραφος 1α, Νεντελτσέβα, ναι, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 1β, τροπολογία 4, Φιλίπ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5, παράγραφος 2, Βαλέσα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6, παράγραφος 2, Τιτσιάνο Μότι. Και εδώ κατά τμήματα, υπέρ για το πρώτο τμήμα κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται, να κάνουμε επαλήθευση, να κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση. Approvo la votazione. Άρχεται η ψηφοφορία. Αν δεν έχετε όλη την κάρτα σα να κάνουμε ψηφοφορία διανατάσσεω χειρό και να μετρήσουμε. Συμφωνείτε? Ωραία. Υπέρ. Και κοντράριο. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7, υπέρ, 14 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 7, παράγραφος 2α, Φιλίπ Μπουλάν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Παράγραφος 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Τροπολογία 9. Keith Taylor υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10 παράγραφος 5 από την υποφινόμενη κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, να επαληθεύσουμε. Για το δεύτερο τμήμα, πάντα διανατάσσεω ισχυρός, Υπέρ. Quindi è approvato con... Εγκρίνεται 12 ψήφοι υπέρ. Κοντράρι. Κατά, ζητώ συγγνώμη. Λέει η Και εσύ Αποχές. Ζητώ συγγνώμη. 12 ψήφοι υπέρ, 5 κατά. Εγκρίνεται. Δεν κάνουμε σωστό έλεγχο. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με να μετράμε λίγο καλύτερα. 12 υπέρ, 6 κατά, εγκρίνεται η τροπολογία. Τροπολογία 11, παράγραφος 5, Keith Taylor και αυτή κατά τμήματα. Υπέρ για το πρώτο τμήμα. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Υπέρ για το δεύτερο τμήμα. Κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Τροπολογία 26, παράγραφος 13α. 12 al paragrafo 5. Τροπολογία 12, παράγραφος 5, κυρία Νεντελτσέβα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13, παράγραφος 5, δεύτερο τμήμα, γέντς, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 14, παράγραφος 5, δεύτερη προστίκη του κυρίου Μότι εδώ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εμενταμέντο 15 al παράγραφο. Τροπολογία 15, παράγραφος 5α 9 του κυρίου Μπουλάν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 16, παράγραφος 7, Βαλέσα, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17, παράγραφος 7α νέα, Νεντελτσέβα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 18, παράγραφος 8, Μότι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 20, παράγραφος 9α, μπουλάν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 21, παράγραφος 9α, νέα, μπουλάν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 22, παράγραφος 10, Νεντελτσέβα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 23, παράγραφος 10α, νέα, Νεντελτσέβα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 24, παράγραφος 11, Μπαλασίτης υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. Τροπολογία 25, παράγραφος 12, γκέντς, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26, παράγραφος 13α, νέα, μπουλάν, υπέρ, κατά, Συγγνώμη, επαναλάβουμε, υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. Ο κύριος Βίλαντ πριν από την τελική ψηφοφορία. Εδώ μπορούμε κάλλιστα να ψηφίσουμε ξεχωριστά, ακόμα και αν δεν είχε αρχικά αποφασιστεί. Δηλαδή το 6 είναι ε, πρώτο και δεύτερο τμήμα υπήρχαν δύο τμήματα και δεν ψηφίσαμε για το δεύτερο, ψηφίσαμε μόνο για το πρώτο. Για το τροπολογία 6. Yes, um, on Πρόεδρε, στην τροπολογία 6 είναι μία τροπολογία, αλλά είχα προτείνει η δεύτερη παράγραφος να ενσωματωθεί σαν ξεχωριστή. Χρειάστηκε λοιπόν να ψηφίσουμε για το σύνολο του κειμένου. Και καταπίπτει, αν κατάλαβα καλά. Academic. Δεν έχει νόημα λοιπόν να επανέλθουμε. Quindi se ho ben capito dobbiamo fare αν κατάλαβα καλά, πρέπει να ψηφίσουμε για την τροπολογία που ε, εισάγει τη δεύτερη παράγραφο, για τη δεύτερο τμήμα, όπως είπε ο κύριος Βίλαντ, πρέπει να κάνουμε και δεύτερη ψηφοφορία. Okay. Διότι εδώ η γραμματεία μου λέει όχι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ξαναψηφίσουμε. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ισχύει. Okay. Ωραία. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Μπορούμε τώρα να ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ομόφωνα εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα την γνωμοδότηση όσου παρουσιάστηκε υπέρ. Υπέρ, κύριε Τσίτσιστερ. Κατά. Αποχές. Και πάλι ομόφωνα εγκρίνεται. Passiamo al punto successivo. Περνάμε στο επόμενο σημείο, γνωμοδότηση επί τη ανακοίνωση σχετικά με την 27η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο τη εφαρμογή του δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση η συγγήτρια η κυρία Άουκεν, στην οποία εδώ το, δίνω το λόγο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που πήρα το λόγο πριν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τους συναδέλφους. Με τους σκιώδεις ηγητές ιδιαίτερα είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση και υπήρχαν κάποια σημεία στα οποία διαφωνήσαμε, ένα συγκεκριμένο σημείο, Πρωτού προχωρήσουμε πάντω στην ψηφοφορία, κυρία Πρόεδρε, ένα πράγμα μόνο θέλω να σα ζητήσω. Με ακούτε, κυρία Ματσόνη, σε εσά μιλάω. Ένα πράγμα θέλω να σα ζητήσω μόνο. Λαμβάνοντα υπόψη ότι ε, η Επιτροπή μα ε, πολλές φορές αντιμετωπίζει το πρόβλημα ότι όταν συνεδριάζει εκτάκτος όπως σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι είναι σε άλλες επιτροπές. Θα πρέπει λοιπόν η ψηφοφορία να γίνεται μία περίοδο που μπορούν και άλλοι συνάδελφοι να είναι εδώ. Δεν αναφέρομαι σε αυτή την ψηφοφορία. Δεν ζητώ κάποια αναβολή αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι θα πρέπει στις επόμενες προφορίες που θα οργανώσουμε να φροντίσουμε ώστε να λαμβάνουν χώρα κάποια στιγμή που μπορούν όλοι οι συνάδελφοι να βρίσκονται εδώ πέρα. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να έχουμε μια πιο, πιο ξεκάθαρη εικόνα της α, πλειοψηφίας στην Επιτροπή αυτή, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να αφαιρθώ τώρα σε δύο προβληματικά σημεία. Τροπολογία 5 που καλύπτει και την 12 τελικά, το ζήτημα αυτό που έχει να κάνει με το δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα. Ελπίζω ότι οι Βρετανοί συντηρητικοί θα είναι υπέρ του να δώσουμε στους πολίτες ευρεία πρόσβαση στα έγγραφα, γιατί αυτό συνάδει πάρα πολύ με αυτά που λένε κατά καιρούς ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε το δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα. Ελπίζω λοιπόν πραγματικά ότι μόνο το ΕΛΚ θα είναι αυτό το οποίο θα αντιταχθεί σε μια τέτοια πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα. Συμφωνώ με την τροπολογία που ζητά καλύτερη πρόσβαση σε όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία είναι ήδη δημόσια, τα οποία έχουν ήδη κοινοποιηθεί. Αυτό είναι σωστό αλλά με ενοχλεί αν στην ε, Επιτροπή αυτή υποστηρίζουμε τους πολίτες θεωρητικά, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε στην ουσία τους πολίτες να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα. Όπως τα ακούσατε χθε στην συζήτηση, η απόφαση αυτή είναι καθαρά πολιτική. Υπάρχει ο κανονισμός 1049, στα πλαίσια του οποίου πρέπει να αποφασιστεί αν θα δώσουμε στους πολίτες μεγαλύτερη πρόσβαση στα έγγραφα. Ελπίζω λοιπόν ότι ε, θα φανεί ότι μόνο το ΕΛΚ αυτό το οποίο φοβάται τελικά τους πολίτες. Αυτό, αυτή είναι η μόνη παρατήρηση που είχα να κάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Άουκεν. Σας ευχαριστούμε και για το έργο σας για το πρώτο έτοιμά σα ε, Θα το εξετάσουμε στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών για την οργάνωση των εργασιών της Επιτροπής μας. Να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την γνωμοδότηση της κυρίας Σάουκεν. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 1 καταπίπτει, τροπολογία 2 παράγραφος 2 της κυρίας Μπασέσκου υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία, συμβαστική τροπολογία 2 παράγραφος 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 3, 4 και 5. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 3, παράγραφος 4, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 6, 7, 8. Τροπολογία 9, παράγραφος 5, της κυρίας Μπασέσκου, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4, παράγραφος 9, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κατά πίπτη 10. Ψηφίζουμε την 11 παράγραφος 13 της κυρίας Μπασέσκου. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 5, παράγραφος 14, υπέρ, κατά, αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Να επαναλάβουμε την ψηφοφορία για τη συμβιβαστική τροπολογία 5 στην παράγραφο 14. Υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία με 13 ψήφους υπέρ. Καταπίπτει η 12. Είμαστε στην τελική ψήφο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ομόφωνα. Να ψηφίσουμε τώρα το σύνολο της γνωμοδότησης υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται ομόφωνα. Ευχαριστούμε. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 15, ετήσια έκθεση για τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών για το 2010 ο εισηγητή είναι ο συνάδελφος Μέγερ, στον οποίο θα δώσω απευθεία το λόγο για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία, διότι μου δίνει τη δυνατότητα να διαρθρώσω αυτό το σχέδιο έκθεσης που έχετε αναχείρας. Έχουμε ήδη λάβει κάποιες τροπολογίες, όλες από την κυρία Μπρέτμαν, και να σας πω ότι σήμερα στις 5 θα γίνει μία συνεδρίαση με τους κοιόδης συγητές όλων των πολιτικών ομάδων προκειμένου από κοινού να επεξεργαστούμε το σχέδιο έκθεσης. Σε άλλες ε, συνεδριάσεις έχουμε παρουσιάσει τις γενικές γραμμές ε, της δομής της έκθεσης. Είναι πλέον έτοιμη και σήμερα το απόγευμα στις 5 θα έχουμε και τη δυνατότητα να ακούσουμε τις προτάσεις από όλους τους κοιόδης εισηγητές των πολιτικών ομάδων, ώστε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, ώστε να καταλήξουμε και στη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση για την έκθεση αυτή. Η έκθεση προσπαθεί, όπως όλες οι εκθέσεις, να αναφέρουν με σαφή τρόπο τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών στη διάρκεια του 2010, κατατάσσοντας τις αναφορές με βάση κάποια κριτήρια, ε, επισημαίνει το ρόλο της Επιτροπής Αναφορών για τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι ασκούν το δικαίωμα της αναφοράς και αναφέρεται ιδιαίτερα στις νομοθετικές αλλαγές που έγιναν μετά από την έναρξη ισχύου της συνθήκη της Λισαβόνας. Οι αναφορές στη διάρκεια του 2010 ε, σας παρουσιάζουμε εδώ κάποια στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των αναφορών, τα θέματα των αναφορών τις ε, χώρες ε, της εθνικότητας των πολιτών που έκαναν περισσότερες αναφορές, η μορφή, ο τρόπος με τον οποίο μας ε, έφτασαν οι αναφορές, είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω επιστολής παραδοσιακά, και επίσης γίνεται και μία ανάλυση όλων των αναφορών, οι οποίες ήταν 1645, υπήρχε μία μείωση της τάξης του 14% σε σχέση με τις περσινές αναφορές αναφέρονται αναφορές, ε, η επεξεργασία που τους έγινε και το αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα των αναφορών. Τα βασικά θέματα των αναφορών ήταν καταρχάς το περιβάλλον, στη συνέχεια τα θεμελιώδη δικαιώματα, η εσωτερική αγορά, δικαιοσύνη, μεταφορές, υγεία, κοινωνικές υποθέσεις, παιδεία, πολιτισμός, ιδιοκτησία και επιστροφές και αποζημιώσεις οι πτυχές που αναφέρονται στην έκθεση έχουν σχέση και με την ίδια την Επιτροπή των Αναφορών υπό την έννοια ότι επισημαίνουμε την ανάγκη να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών σε αυτή τη διαδικασία λήψης απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σημασία και το δικαίωμα του να καταθέσει κάποιος αναφορά τη σχέση της Επιτροπής Αναφορών με άλλες ε, επιτροπές ε, του Κοινοβουλίου, είναι, που είναι ένα θέμα που συζητάμε στην Επιτροπή μας ε, στη διάρκεια αυτής της θητείας, το ρόλο της Επιτροπής μας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ανάγκη, όπως ζητήθηκε και στην ετήσια έκθεση που παρουσίασε ο κύριος ιτουργάιθ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δίνει τακτικά πληροφορίες για το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι διαδικασίες, ε, ένα παράρτημα για την Επιτροπή Αναφορών και τη σχέση με το Συμβούλιο της Ευρώπης, μία παράγραφο για την Επιτροπή Αναφορών και τον ε, Συνήγορο του Πολίτη. Η Επιτροπή Αναφορών και η σχέση της με τους Ευρωπαίους πολίτες, οι ανακοινώσεις για τα θέματα του περιβάλλοντος που ανησυχούν ε, περισσότερο την Επιτροπή μας. όσον αφορά το κοινοτικό δίκαιο, την ε, η πρωτοβουλία των πολιτών, τα θεμελιώδη δικαιώματα και κατόπιν γίνεται μια και περιγραφή των αποστολών που κάναμε στη διάρκεια του 2010. Επισημαίνουμε τις πιο σημαντικές όπως ήταν αυτή στην Ουέλβα, ε, στην ε, Καμπανία στην Ιταλία, στην Αυστρία και αναφέρουμε συνοπτικά τα συμπεράσματα. Θα ήθελα κυρίες και κύριοι να σας επαναλάβω ότι πέραν των παρεμβάσεών σα, σήμερα το απόγευμα στι 5 θα έχουμε μια συνεδρίαση με του συντονιστέ για να, με του κοιόδης ηγητές, για να ολοκληρώσουμε τι θέσει όλων των πολιτικών ομάδων με διάθεση όπω πάντα σε αυτή τη μορφή τη εκθέσεις να υπάρχει η μέγιστη δυνατή συνένεση των μελών τη Επιτροπή. Ε, προθεσμία και κατάθεση τροπολογιών 26 Μαΐου στις 3 ε, και ελπίζω μετά και από την απογευματική συνεδρίαση να δώσουμε το πράσινο φως και να παρουσιάσουμε σε μια μελλοντική συνεδρία της Επιτροπής μας το σύνολο της έκθεσης οριστικοποιημένο στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μέγερ για την ε, παρουσίασή του μας έδωσε και τις προθεσμίες για την κατάθεση τροπολογιών και τη συζήτηση αυτής της έκθεσης, η οποία θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Ιουνίου. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Γιάρχης. Äh, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κυρίως γιατί θα συναντηθούμε σήμερα το απόγευμα και θα μιλήσουμε για την έκθεση. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και η ετήσια έκθεση πιστεύω θα πρέπει να υποστηριχθεί με μεγάλη πλειοψηφία εδώ στην Επιτροπή. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω, θα τις επαναλάβω και σήμερα το απόγευμα. Πιστεύω ότι όσον αφορά τις αναφορές οι οποίες ε, αφορούν υποθέσεις που εκκρεμούν ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα πρέπει να έχουμε μια ειδική διατύπωση. Ο καθένας μπορεί εδώ να εκφράσει την επιθυμία του να κάνει κάτι η Επιτροπή Αναφορών για αυτές τις αναφορές. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε τίποτα εφόσον εκκρεμεί η υπόθεση και δεν υπάρχει απόφαση. Δεύτερον, έχω κάποιες προτάσεις που θέλω να κάνω. Ξέρετε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρω το θέμα αυτόν, αλλά θα τις κάνω πολύ συγκεκριμένα σήμερα το απόγευμα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Μέιερ για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Το σχέδιο αυτό έκθεσης επιβεβαιώνει κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι. Η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Αναφορών, αποτελεί το πιο, την πιο δραστήρια διεπαφή, αν θέλετε, ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, την, και τους Ευρωπαίους πολίτες. Επίσης, με τις συνθήκες της Λισαβόνας έχουν αυξηθεί οι αρμοδιότητες αυτές που έχει η Επιτροπή μας. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να υπογραμμίζει τις προσπάθειες που καταβάλουν όλοι οι συνάδελφοι προκειμένου να ενδυναμωθεί η συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους προσώπους των πολιτών και προκειμένου να βρεθεί πάντα ένα συμβασμός και να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις. Ω προ το περιεχόμενο τώρα τη έκθεση πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση, ε, βάσει τη οποία θα υποβάλω και δύο τροπολογίε. Είναι σαφέ ότι αντιμετωπίσουμε πάντα ένα σημαντικό πρόβλημα. Το ότι δεν αντιδρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάρα πολύ γρήγορα, ιδίω όσον αφορά τι αναφορέ εκείνε που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Αν δεν δημιουργηθούν συγκεκριμένε προθεσμίες, αν δεν δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, κάθε φορά που υποβάλλεται μια τέτοια αναφορά, ένα πρόγραμμα πιεστικό για τα κράτη-μέλη, τελικά δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα και δεν θα μπορούμε σε καμία περίπτωση να εμποδίσουμε την ε, καταστροφή του περιβάλλοντος. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση και η Επιτροπή μας πρέπει να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεύτερη παρατήρηση, η σχέση που έχουμε εμεί ω Επιτροπή με τα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή Αναφορών έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τα κράτη-μέλη, μια ξεχωριστή σχέση με τα κράτη-μέλη. Βλέπουμε όμω ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα κράτη-μέλη τα οποία αδιαφορούν ή πολλέ φορέ ακόμα και περίφρονούν τη δραστηριότητα τη Επιτροπή Αναφορών. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί στο μέλλον. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να το αποδεχόμαστε. Πρέπει να θέσουμε ένα τέρμα στην στάση αυτή. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα μηχανισμό που θα μας επιτρέψει να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να απαντούν γρήγορα κάθε φορά που υποβάλλεται μία αναφορά. Χρειαζόμαστε μια γρήγορη και κατάλληλη απάντηση. Εμεί είμαστε άλλωστε εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών, σε εμά απευθύνονται κάθε φορά που καταθέτουν μια αναφορά. Πάρα πολλέ φορέ λάβαμε απαντήσει, οι οποίε ήταν ιδιαίτερα επιφανειακέ, πολλέ φορέ ακόμα και προσβλητικέ για την Επιτροπή μα. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ και στο ότι ε, η Επιτροπή μας και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, καθώς επίσης και η Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων, έχουν ήδη αρχίσει να επεξεργάζονται την εξής ιδέα, να δημιουργηθεί ένας ε, μηχανισμός, ο οποίος θα επιτρέπει να δημιουργηθεί μία νομοθεσία η οποία θα υποχρεώνει ουσιαστικά τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμορφώνονται με τις δικές μας τις αποφάσεις. Είδαμε πολλές φορές ότι οι ίδιες οι διατάξεις της χάρτας παραβιάζονται και ακόμα και στις περιπτώσεις αυτές οι ε, απαντήσεις που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαίτερα δειλές ιδιαίτερα ήπιες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα λέει ότι δεν υπάρχουν νομικά μέσα, δεν υπάρχουν νομικέ ικανότητε, δυνατότητε προκειμένου να διορθωθεί η κατάσταση κάθε φορά που υπάρχει μια καταγγελία, μια αναφορά. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι δική μα υποχρέωση να, έχουμε μία, να ξεκινήσουμε μια κοινή προσπάθεια προκειμένου να δημιουργηθεί ο κατάλληλο νομοθετικό μηχανισμό που θα επιτρέπει την ε, εφαρμογή, την πραγματική υλοποίηση τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και που επιτέλου θα καλούμε τα κράτη-μέλη να συμμορφώνονται με την κοινοτική αυτή νομοθεσία και να μην τη θεωρούν απλώς πολιτική δήλωση. Δείτε για παράδειγμα τις α, τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή τα ανθρώπινα δικαιώματα ή πολλές άλλες θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, οι οποίες πολύ συχνά δεν αντιμετωπίζονται με τον κατάλληλο τρόπο από τα κράτη-μέλη. Πρέπει να σταματήσει η τάση αυτή, πρέπει να διορθωθεί η κατάσταση. Είναι, δική μας, είναι δικό μας καθήκον ως Επιτροπή Αναφορών να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό και είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σε ευχαριστήσω για την έκθεση αυτή και να κάνω μια παρατήρηση όσον αφορά τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη και το ότι τα κράτη-μέλη πολλές φορές δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας, δεν θα πρέπει ίσως να κατονομάσουμε αυτές τις χώρες, προκειμένου να ασκηθεί κατά αυτόν τον τρόπο πίεση στα εν λόγω κράτη-μέλη, προκειμένου να επέλθει τελικά η ευκταία αυτή αλλαγή που θέλουμε στη στάση τους. Σαφώς θα πρέπει να υπάρχει ένα κατάλληλο κλίμα συνεργασίας με τα κράτη-μέλη. Το έχουμε επαναλάβει πάρα πολλές φορές αυτό στο παρελθόν. Η κυρία Όκεν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω κι εγώ, όπως και άλλοι συνάδελφοι, στην μητρική μου γλώσσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή Έρχεται την κατάλληλη στιγμή η έκθεση αυτή. Αναφέρεται σε πολύ κέρια ζητήματα για την Επιτροπή μα. Ήδη χθε μιλήσαμε για κάποια από τα ζητήματα αυτά. Αναφερθήκαμε στο ρόλο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, αναφερθήκαμε σε κάποια προβλήματα τα οποία προκύπτουν, προβλήματα τα οποία είναι πολύ πιο πολιτικά και όχι τόσο νομοθετικά. Πολλές φορές ακολουθείται μία πάγια πολιτική παράδοση και βλέπουμε ότι αυτή οδηγεί σε πολλές καθυστερήσεις ή σε πολλά εμπόδια όσον αφορά την επίλυση κάποιων προβλημάτων. Μόλον ότι πολλές φορές ακολουθεί τη διαδικασία επί παραβάση, υπάρχουν ε, υποθέσεις οι οποίες δεν επιλύονται εύκολα, ακριβώς επειδή η πρόσβαση προβληματων μολονοτι οτι πολλες φορες ακολουθει τη έγγραφα δεν είναι αυτή που θα πρέπει να ήταν. Υπάρχει γενικότερα μια πρόσβαση στα έγγραφα και ιδίω μέσω του διαδικτύου και στην έκθεσή μου Μάλλον για την έκθεση αυτή έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες που έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτό το πράγμα, τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα. Θα πρέπει όλα αυτά τα έγγραφα να είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο προκειμένου να γνωρίζουμε ακριβώς πώ έχει κατάσταση για κάθε αναφορά. Σαφώς θα πρέπει να σεβαστούμε τα όσα λέγονται στον κανονισμό 1049, αλλά από την άλλη είναι εξίσου σημαντικό να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη πρόσβαση σε όλα αυτά τα έγγραφα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει, σε ποια σημεία μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, όπως ακριβώς είπε και ο συνάδελφος Μέιερ πριν από λίγο. Όσο θα υφίστανται τα προβλήματα αυτά, οι πολίτε δεν θα μα παίρνουν σοβαρά, τα κράτη-μέλη δεν θα ανταποκρίνονται στι εκκλήσει μα και δεν θα καταφέρνουμε να επιλύουμε σημαντικά προβλήματα όπω αυτά που έχουν να κάνουν με την καταστροφή του περιβάλλοντο. Πιστεύω ότι πρέπει να επιμείνουμε σε όλα αυτά τα σημεία. Μαζί με του σκιώδει εισηγητέ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε κάποια εκκρεμή προβλήματα προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Θα ήθελα να αφαιρθώ στο σημείο S, στο σχέδιο αυτό έκθεση. Σε αυτό το σημείο λέγεται ότι θα πρέπει να ενημερωνόμαστε κατά τακτική βάση για τόσα συμβαίνουν. Μου προκαλεί εντύπωση το ότι δεν μας ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάποιες διαδικασίες, ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία με τις δημόσιες προμήθειες στην Ισπανία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μας είχαν δοθεί πολύ περισσότερες πληροφορίες για το ζήτημα αυτό. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο Φίλιπ Μέιερ, συμφωνώ με τα όσα είπε και ο Βικτόρ. Τα ζητήματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και ουσιαστικά θα βελτιώσουν την λειτουργία της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ τους αδέλφους Ο κύριος Φλόιντ, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν θέλει να λάβει το λόγο. Έχει το λόγο. Μας ικανοποιεί η έκθεση αυτή, φορά του 25-26. Πιστεύω ότι αντιστοιχεί στη συζήτηση που είχαμε στην Ολομέλεια πέρσι. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι. Παράγραφος 13. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου είναι αυτή η οποία έχει συντάξει τις κατευθυντήριες γραμμές και υπάρχουν και κάποιες προτάσεις τις οποίες θέλω να υποβάλω. Είναι μάλλον συντακτικές πριν την συνάντηση των σκιώδων εισηγητών σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Φλόιντ. ο κύριος Μάγερς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας, οι οποίες ε, θέλουν να βελτιώσουν το κείμενο. Ελπίζω οι προτάσεις αυτές, οι οποίες είναι ήδη αποδεκτόες να μπορέσουν σήμερα το απόγευμα να βρουν και την ανάλογη διατύπωση για να συμπεριληφθούν στο κείμενο. Ο κύριος Γιάρ έχει δίκιο στην πρώτη παρέμβαση που έκανε για το γεγονός ότι έχουμε και αρμοδιότητες που έχουν σχέση και με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εδώ υπάρχει και μία σύγκρουση ε, πολιτικού και δικαστικού ε, κλάδο και πρέπει να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές άγουσες, τις οποίες πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη. Όσον αφορά τώρα τις νέες αναφορές και το πώς πρέπει να τις ε, προχωρούμε, νομίζω ότι ο κύριος Γιάρου ούτως ή άλλως σήμερα το απόγευμα θα μπορέσει σε διευκρινίσει τι εννοεί και να το συμπεριλάβουμε στο κείμενο. Ο κύριος Μποστινάρου ε, πάντα κάνει σωστές εκτιμήσεις. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ιδιαίτερη επιτροπή. Η Επιτροπή Αναφορών είναι αυτή η οποία έρχεται σε άμεση επαφή με τους Ευρωπαίους πολίτες και είναι ιδιαίτερη και η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την οικονομία και το μοντέλο της ευημερία και αυτή η σχέση με τους πολίτες είναι μια πολύ ειδική σχέση συμφωνώ ότι θα πρέπει να επισημάνουμε το, η μέθοδο εργασίας της, Ευρω... της Επιτροπής μας, διότι πάντα εδώ τα μέλη της Επιτροπής προσπαθούν να καταλήξουν σε συνένεση. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο εμφανίζεται συνεχώς σε όλες τις εκθέσεις και υπάρχει και το πρόβλημα με την παρουσίαση μιας, επιτρο... μιας αναφοράς που έχει σχέση με το περιβάλλον και το γεγονός ότι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθυστερούν και η απάντηση έρχεται πολύ καθυστερημένη και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφεύγουμε αυτά που μπορούμε να αποφύγουμε. Πάντα προσπαθούμε να περιορίσουμε τα χρονικά περιφέρεια και να βρίσκουμε λύση νωρίτερα. Αυτό ανέφερε και η κυρία Βέρτμαν. Η σχέση που έχουμε ως Επιτροπή με τα κράτη-μέλη είναι σημαντική πρόκειται για μια σχέση η οποία καθορίζεται ε, δυστυχώς όχι μέσω συνεργασίας, αλλά υπάρχει μια απόσταση και θα πρέπει να ομολοποιήσουμε τις σχέσεις ε, μεταξύ Επιτροπής Αναφορών και κρατών μελών όταν ε, μια αναφορά άπτεται ενός συγκεκριμένου κράτους. Ε, και η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων πράγματι δεν θα πρέπει να είναι ένας πολιτικός χάρτης, αλλά ένας χάρτης ο οποίος θα έχει και νομοθετικές πτυχές από πλευρά μου έχετε όλη την υποστήριξη ώστε να το επιτύχουμε αυτό και να έχουμε και μεγαλύτερη βαρύτητα για τη χάρτα. Να ευχαριστήσω την κυρία Βάρτμαν για τα σχόλιά της και για το γραπτό κείμενο που μου έχει δώσει και στην κυρία Άουκεν να πω ότι πράγματι στο σημείο S που αναφερόμαστε στην ανάγκη να προχωρούν όλες οι διαδικασίες ομαλά, νομίζω ότι θα πρέπει να προσθέσουμε ότι και η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα βάσει του ε, κανονισμού 1049 όντως είναι απαραίτητη. Νομίζω ότι σήμερα το απόγευμα θα μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε το σχέδιο έκθεσης ώστε να το παρουσιάσουμε από εκεί και πέρα ως έκθεση με τη συνένεση όλων των μελών της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Μέγερ. Σας υπενθυμίζω η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι 26 Μαΐου στις 3 το απόγευμα και η έκθεση στη συνέχεια θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας τον Ιούνιο. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, σημείο του 16, δύο αναφορές που θα συζητηθούν από κοινού, η 475 του 2010 από τον Αλμπέρτο Παθ Βίνιας για τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών των δικαιωμάτων και η 1326 του 2010 του Τσιπριάνο Ρικάρντο Λούστρε Μαρτίνεθ και πάλι Ισπανική Ιθαγένεια, εξ ονόματο τη Ένωση Long Hope, σχετικά με την κατάσταση των Ισπανών ναυτικών οι οποίοι εργάζονται ω μέλη του πληρώματο σε σκάφη που φέρνει την Ορβηγική σημαία. Είναι παρόν ο δεύτερος ε, αναφέρον και του δίνω το λόγο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Σα ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τα αιτήματά μα εδώ. Είμαστε ένα σύλλογο πρώην Ισπανών ναυτικών που εργάζονταν σε νορβηγικά σκάφη με έδρα στη Γαλλικία, μια ε, αλλιευτική περιοχή και παρουσιάζουμε το αίτημά μας στην αναφορά αυτή διότι δεν αναγνωρίζονται τα εργασιακά μας δικαιώματα στην Νορβηγία διότι βάσει της νομοθεσίας της Νορβηγίας τότε δεν θεωρούμασταν κάτοικοι της Νορβηγίας διότι εργαζόμασταν ε, σε ανοιχτή θάλασσα. Από το 1963 υπάρχει μία σύμβαση για να μην υπάρχει ε, διπλή φορολόγηση. Βάσει αυτού οι ναυτικοί οι οποίοι παρήχαν υπηρεσίε σε νορβηγικές επιχειρήσεις έπρεπε να θεωρούνται για φορολογικούς σκοπούς μη κάτοικοι. Παρά το γεγονός ότι η διοίκηση της Νορβηγίας έκανε κρατήσεις ε, ίδιες με οποιονδήποτε άλλο εργαζόμενο. Αναγνώριζε ρητός λοιπόν ε, τους Ισπανούς ναυτικούς ως μόνιμους κατοίκους. Το ίδιο πρόβλημα συνέβη και με τους Ισπανούς εργαζομένους στη Δανία, η οποία είναι χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν τέλει αναγνώρισε ότι υπάρχει διάκριση στη διαδικασία και αναζήτησε μία ε, λύση για τους ε, εργαζομένους που πλήττονταν ζητάμε αναγνώριση των ετών εργασίας στα νορβηγικά σκάφη και να ε, δοθούν τα συντεξιοδοτικά δικαιώματα και να ε, ε, καλυφθούμε από το κοινωνικό σύστημα. Ζητάμε από την ορφαγική κυβέρνηση την αποζημίωση των ποσών που παρακρατήθηκαν και να δοθούν σε ένα εφάπαξ ποσό με αναλογία στα σημερινά ε, δεδομένα, οικονομικά δεδομένα και επειδή είμαστε Ευρωπαίοι εργαζόμενοι ζητάμε την υποστήριξη των πολιτικών ομάδων ώστε οι εργαζόμενοι από διάφορα κράτη-μέλη, όχι μόνο Ισπανία αλλά και Πορτογάλοι, Ιταλοί, Γερμανοί, Βέλγοι και όλοι να μην ε, είναι αντικείμενο διάκρισης ε, στις κοινωνικές τους ασφαλίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ ο λόγος στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Βορύδης. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια δύσκολη κατάσταση, μια κοινωνική αδικία. Γιατί δημιουργήθηκε αυτή η άδικη κατάσταση. Καταρχήν το κοινοτικό δίκαιο δεν ίσχυε πριν το 1994 στην Νορβηγία. Μόνο το, η εθνική νομοθεσία ήταν σε ισχύ. Η νομοθεσία της Νορβηγίας προβλέπει την ε, κατοικία στο έδαφος της χώρας για να αναγνωριστούν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Παραδείγματος χάρη, ένα άτομο που εργαζόταν σε πλατφόρμα εξόριξης πετρελαίου δεν μπορούσαν να καλυφθούν από τα συνταξιοδοτικά ταμεία ε, στην Νορβηγία και απλώς καλύπτονταν η ιατρική τους περίθαλψη σε περίπτωση ατυχημάτων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι αρμόδια και δεν ε, έχει νομικά εργαλεία έτσι ώστε να ζητήσει από την ε, Νορβηγία αναδρομικά την κάλυψη αυτών των εργαζομένων. Παρ' όλα αυτά, ο κανονισμός 883 του 2004 που προβλέπει τις περιπτώσεις αυτές δίνει το δικαίωμα στις αρχές των χωρών αυτών να συνάψουν διμερείς συμφωνίες προς όφελος των εργαζόμενων αυτών. Για να υπάρξει λοιπόν κοινωνική δικαιοσύνη, οι αρμόδιες αρχές της Ισπανίας και της Νορβηγίας θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή έτσι ώστε να συναυθεί μια τέτοια διμερή συμφωνία προς όφελος και προς συμφέρον των εργαζόμενων αυτών. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να δώσω και μια άλλη πληροφορία η οποία μπορεί να είναι χρήσιμη για αυτήν την αναφορά. Το δικαστήριο θα αποφανθεί όσον αφορά την ισχύ του κοινοτικού δικαίου, την εφαρμογή του ε, κοινοτικού δικαίου στις πλατφόρμες εξόρεξης που βρίσκονται κοντά στις ακτές της Ολλανδίας. Πρόκειται για την υπόθεση 4710 του 2006. Πρόκειται για έναν εργαζόμενο ο οποίος εργαζόταν στις πλατφόρμες εξόρυξης, δεν κατοικούσε όμως στην Ολλανδία, άρα δεν μπορούσε να καλυφθεί από τα συνταξιοδοτικά ταμεία της Ολλανδίας. Ήταν Ισπανός. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται και εάν είναι θετική, πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να υπάρξει μία συμφωνία μεταξύ Ισπανίας και Νορβηγίας για τους εργαζόμενους αυτούς οι οποίοι εργαζόταν σε σκάφη ή πλατφόρμες ε, νορβηγικές. Επαναλαμβάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αρμόδια και δεν έχει κανένα νομικό εργαλείο έτσι ώστε να αναγκάσει την Νορβηγία. Θα κάνει όμως ό,τι μπορεί έτσι ώστε να ενθαρρύνει τις δύο αυτές χώρες, την Ισπανία και την Νορβηγία, έτσι ώστε να βρεθεί μια δίκαιη λύση στο πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ για τη συνεργασία και την ε, διαθεσιμότητά σας, ο κύριος Ιτουρκάης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρα. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο συμβαίνει επειδή δεν είναι συντονισμένες οι νομοθεσίες ε, διαφόρων κρατών και δυστυχώς ε, δυσχεραίνουν ιδιαίτερα τη ζωή ενός πολίτη. Όταν φτάνει λοιπόν ε, η ηλικία συνταξιοδότησης αυτών των Ισπανών εργαζομένων, η νορβηγική κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματά τους και ενώ η Ισπανική κυβέρνηση δεν μπορεί να τους αναγνωρίσει ε, συνταξιοδοτικά δικαιώματα ζητά να τους αναγνωριστούν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στη χώρα που είχαν μεταναστεύσει, δηλαδή στην Νορβηγία. Ακούσαμε όμως τους ίδιους τους ναυτικούς εδώ και υπάρχει ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να δημιουργηθούν ερωτηματικά. Όσο και αν σεβόμαστε την Νορβηγική νομοθεσία, κυρία Πρόεδρε, είναι εκπληκτικό από νομοθετικής πλευράς το γεγονός ότι η Νορβηγία δεν δίνει καθεστώς μόνιμου κατοίκου σε Ισπανούς ναυτικούς οι οποίοι πέρασαν όλη τους τη ζωή εργαζόμενοι σε νορβηγικά σκάφη με νορβηγική σημαία βάσει νορβηγικής νομοθεσίας και καταβάλλοντας και φόρους ε, στην ε, νορβηγική ε, εφορία. Η νορβηγική κυβέρνηση λοιπόν θα τους αναγνώριζε φορολογική νορβηγική κατοικία, αλλά δεν τους αναγνωρίζει μόνιμη κατοικία στην Νορβηγία όταν πρέπει να τους καταβληθούν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Ένα από τα βασικά δικαιώματα των κοινωνικών και δημοκρατικών κρατών ε, του 20ου αιώνα είναι να φροντίζουμε τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών και να τους δίνονται τα δικαιώματα αυτά σε κάθε περίπτωση ε, η οποία μπορούσε να δημιουργήσει αμφισβήτηση και ανισότητα μεταξύ ίσων ε, λόγω συγκεκριμένων συνθήκων. Δεν θα πρέπει να πλήττονται τα δικαιώματα των πολιτών σε καμία περίπτωση. Όλα αυτά τα είπα διότι γίνεται μια κατάφορη αδικία εδώ και εγώ νομίζω ότι θα μπορούσα να πάω και λίγο περαιτέρω το θέμα. Ουσιαστικά τους καταλυστεύουμε αυτούς τους ανθρώπους, δεν έχουν πλέον δικαιώματα διότι υπάρχει αυτό που έλεγε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των ναυτικών αυτών, κατά των ανθρώπων αυτών, υπάρχει μια μεγάλη, πολύ σοβαρή ανευθυνότητα, η οποία είναι γνωστή τη πάση και όλοι απλώς σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και λέμε πράγματι είναι παρατυπή αυτό που συμβαίνει, είναι αδικία αυτό που σας συμβαίνει, αλλά κύριε και κύριοι δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όχι, δεν είναι έτσι. Πρέπει να αναζητήσουμε λύση. Είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε λύση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσει να διαφυλάξει τα δικαιώματα των εργαζομένων και θα πρέπει να αναζητήσει έναν τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι αυτοί να μην μείνουν ανυπεράσπιστοι. Διότι ήδη μας το λέει ότι είναι ανυπεράσπιστη αυτή τη στιγμή και αυτό που ζητώ είναι να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε μαζί με την κυρία Πρόεδρο να αφήσουμε την αναφορά ανοιχτή, να μην κλείσει το ζήτημα και όπως σας έλεγα προηγουμένως να προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση. Μία λύση που θα δικαιώσει όλους αυτούς τους πολίτες που δεν έχει σημασία αν είναι Ισπανοί οι πολίτες ή πολίτες οποιασδήποτε άλλη χώρας, τους ε, καταπατούνται τα δικαιώματά τους. Το αναγνωρίζει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σάντσες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω τους αναφέροντες από τη Γαλλικία, διότι είναι και η δικιά μου η περιφέρεια, να εκφράσω την αλληλεγγύη και να πω ότι πρέπει να προασπίζονται τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Εργάζονταν υπό νορβηγική σημαία σε εγκαταστάσεις της Νορβηγίας, κατέβαλαν τους φόρους τους και το κοινωνικό σύστημα της Νορβηγίας χρηματοδοτείται μέσω της φορολογίας και επομένως θα πρέπει να αποπληρώνονται βάσει μια σύμφασης ε, του 1964 που τους θεωρεί μονίμους κατοίκους. Το 2008 είχαμε και μία ερώτηση στην οποία απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του θέματος, ε, ζήτησε πληροφορίες, οι πληροφορίες αυτές ε, συγκεντρώθηκαν και το 2010 αυτή τη στιγμή συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες, εγώ παρουσίασα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακόμα δεν έχω λάβει απάντηση δεν είμαι πολύ ικανοποιημένο ε, από το γεγονός ε, και μόνον ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα κοινωνικής δικαιοσύνης και ούτε θα είμαι ικανοποιημένο από το όσα μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν είναι της αρμοδιότητάς τους. Η απάντησή μου στην ερώτησή μου του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου είπε ότι βάση του κανονισμού σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης είναι προφανές ότι βάσει του άρθρου 94.2 του συγκεκριμένου κανονισμού θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις εισφορές οι οποίες καταβλήθηκαν ή θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί στην περίοδο πριν από την ένταξη στη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και του χώρου ΕΟΧ της Νορβηγίας και θα πρέπει να συνάθουν τα πάντα με τον κανονισμό. Δεύτερον, Υπάρχει το άρθρο 87.4 του νέου κανονισμού, το οποίο απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι τα δικαιώματα θα πρέπει να ε, καταβληθούν εφάπαξ. Και τα δύο θέματα λοιπόν αφορούν την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακα των συνθήκων θα πρέπει να φροντίσει να τηρούνται απολύτω οι όροι. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθήσει να διορθώσει αυτή την αδικία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει τις σχέσεις ώστε να τηρηθεί συμφωνία, να υπάρξει μια συμφωνία η οποία θα μπορούσε να είναι και διμερής, αλλά κατά την άποψή μου θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, διότι μπορεί να υπάρχουν ανάλογες περιπτώσεις σε άλλα κράτη-μέλη τα οποία χρήζουν τις ίδιες λύσεις και επίσης θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκός κανονισμός επί του θέματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εκφράσει την αλληλεγγύη της όχι μόνο με λόγια, αλλά να υλοποιήσει τη δέσμευσή της, να καλέσει την Ορβηγία και την Ισπανία να βρουν ε, μία λύση ε, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και το θέμα αυτό να μείνει ανοιχτό μέχρι να βρούμε την κατάλληλη λύση. Ευχαριστώ. Muchas gracias, señora presidenta. Yo también he venido aquí para... Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα Καταρχήν να σας πω ότι θα ήθελα να υπερασπιστώ αυτούς τους Ισπανούς ναυτικούς οι οποίοι εργάστηκαν τη δεκαετία του 70, 80 και 90 σε νορβηγικά σκάφη. Γνωρίζω πολύ καλά την περίπτωση αυτή και εδώ και χρόνια έχω επαφές ε, με τον πρόεδρο του συλλόγου αυτού που συγκεντρώνει όλους αυτούς τους ναυτικούς. Πέρσι είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό πώς θα μπορούσαν δηλαδή να συντονιστούν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Προσπαθούμε να βρούμε μία λύση από κοινού με την Επιτροπή για αυτά τα πολύ περίπλοκα θέματα. Οι ναυτικοί αυτοί βρίσκονται σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση και η Ισπανία δεν αναγνωρίζει την εργασία του στην Νορβηγία, η δεν Νορβηγία δεν θεωρεί ότι πρέπει να τις καταβάλει συνταξιοδοτικά δικαιώματα, καθότι δεν ήταν μόνιμοι κάτοικοι και δεν μπόρεσαν να συνεισφέρουν ε, στο σύστημα το νορβηγικό. Παρόλα αυτά, όπως ακούσατε, πλήρωναν φόρους, αρκετά υψηλούς φόρους ε, στην Νορβηγία η ναυτική αυτή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω λάβει στην Νορβηγία, η κοινωνική εισφορά κυρίως χρηματοδοτείται από τη φορολογία και όχι μόνο από τις ε, εισφορές των εργαζομένων. Η φορολογία λοιπόν έχει καταβληθεί από τους ναυτικούς αυτούς. Μήπως θα πρέπει λοιπόν τουλάχιστον να τους αποζημιωθεί ο φόρος που κατέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια, αφού είναι σήμερα γνωστό ότι το κοινωνικό σύστημα στην Νορβηγία χρηματοδοτείται από την φορολογία. Η Επιτροπή μας λέει ότι δεν είναι αρμόδια. Θα ήθελα παρόλα αυτά να πω ότι ακόμα και αν η Νορβηγία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση για τους εργαζομένους της Ισπανίας και άλλων χωρών εξάλλου, γιατί δεν αφορά μόνο την Ισπανία το θέμα αυτό. Επιμένω ότι η Επιτροπή πρέπει να παίξει έναν πιο ενεργητικό ρόλο, πιο αποτελεσματικό ρόλο. Να προσπαθήσετε να δείτε, παραδείγματο χάρη, τι ποσά καταβλήθηκαν μέσω των φόρων και να δούμε αν μπορεί ένα τμήμα αυτών των ποσών να επιστραφεί στους εργαζόμενους από τη στιγμή που δεν έχουν δικαιώματα. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει όσον αφορά τις προσπάθειές της και να παρακολουθήσουμε όλοι την κατάσταση και βεβαίως περιμένουμε με ανυπομονησία και την απόφαση του δικαστηρίου γιατί αυτό αφορά και άλλους εργαζόμενους όπως τους Ολλανδούς. Επαναλαμβάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και η Επιτροπή μας θα πρέπει να συνεχίζουν να παίζουν έναν ενεργό ρόλο και να παρακολουθήσουμε τι γίνεται με τους εργαζόμενους αυτούς οι οποίοι πραγματικά έχουν συνεισφέρει στο σύστημα της Νορβηγίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση και στους αναφέροντες αλλά και στην Επιτροπή. Υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο όσον αφορά τις ε, εισφορές σας ε, στο νορβηγικό σύστημα, τη φορολογία δηλαδή που πληρώνετε. Αν ναι, κατά την άποψή μου, είναι προφανές ότι οι αναφέροντες θα πρέπει να λάβουν κάποια ποσά, να τους επιστραφούν κάποια ποσά. Αυτό είναι για μένα θέμα ε, δικαιοσύνης. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχουν συνεισφέρει στο σύστημα και δεν έχουν πάρει τίποτα, θα πρέπει τα ποσά αυτά να τους επιστραφούν. Νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που υπάρχει στο ευρωπαϊκό δίκαιο, από τη στιγμή δηλαδή που έχουν πληρώσει στο νορβηγικό σύστημα και δεν τους επιστρέφεται τίποτα μέσω των συνταξιοδοτικών ταμείων. Έχω την εντύπωση ότι εδώ πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν παραβιάζονται οι αρχές του κοινοτικού δικαίου και η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει το θέμα αυτό. Δεν νομίζω ότι αφορά μόνο την Ισπανία εξάλλου η υπόθεση αυτή. Σαν ε, Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να κάνουμε ένα διάβημα προς την Ορβηγική κυβέρνηση να γράψουμε στον διαμεσολαβητή. Είναι αδύνατο να δεχτούμε. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Δεν το πιστεύω ότι μπορούμε να δεχτούμε μια τέτοια κατάσταση στην Ευρώπη σήμερα. Η Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να επιμείνει. Και ήδη από το 1994 γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Δεν έχει βρεθεί λύση. Από τη στιγμή που κάποιος έχει εργαστεί, έχει συνεισφέρει σε ένα σύστημα κοινωνικών παροχών, δεν μπορεί να μην παίρνει τίποτα σε αντάλλαγμα. Θα ήθελα λοιπόν να έρθουμε σε επαφή με τις νορβηγικές αρχές, να πιέσουμε έτσι ώστε να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Ευρώπης και Νορβηγίας, αν όχι διμερείς μεταξύ Ισπανίας και Νορβηγίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ο κύριος Μάγερ. Θα ήθελα να σας πω και εγώ θεωρώ την υπόθεση αυτή απαράδεκτη. Στηρίζουμε αυτούς τους ε, Ισπανούς ναυτικούς και βεβαίως βάση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δεν είναι δυνατόν κάποιος να έχει συνεισφέρει σε ένα κοινωνικό σύστημα και να μην παίρνει τίποτα σε αντάλλαγμα. Θα πρέπει βεβαίως να βρεθεί μια λύση. Συμφωνώ απολύτως με όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο μέχρι τώρα. Με όλους. Και θεωρώ και εγώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι πολύ πιο απαιτητική έχει αρμοδιότητες. Προτείνω λοιπόν η Επιτροπή να είναι πιο απαιτητική, αλλά και εμείς σαν Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση και να αποταθεί τη στιγμή στις Ισπανικές αλλά και στις Νορβηγικές αρχές έτσι ώστε να συναυθεί μια συμφωνία. Ο διαμεσολαβητής επίσης μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Στην ετήσια έκθεση είδαμε τι μπορεί να αποφέρει η παρέμβασή του και όπως είπε και η Επιτροπή μπορούμε να ζητήσουμε και στις δύο ενδιαφερόμενες χώρες μέσω μιας διμερούς συμφωνίας να αναγνωριστούν τα δικαιώματα αυτών των εργαζομένων. Η Νορβηγία θα πρέπει εδώ να αναλάβει τις ευθύνες της. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι σαφές ότι έχουμε μια ξεκάθαρη υπόθεση εδώ μπροστά μας. Βλέπουμε ότι de jure και de facto τα πράγματα διαφέρουν πάρα πολύ. Γιατί βλέπουμε ότι ενώ υπάρχει μια εργασιακή σύμβαση και απαιτείται από τους ναυτικούς να καταβάλουν φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλειας στον νορβηγικό προπολογισμό, de facto τους ε, αντιμετωπίζουν ως διαμένοντες πολίτες της Νορβηγίας. Όταν ε, καταβάλει κανείς φόρους όμως, θα πρέπει να τον αγνωρίζονται και δικαιώματα. Όταν έρχεται η στιγμή της σύνταξης βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί δεν αντιμετωπίστηκαν ούτε ως πολίτες, ούτε ως κάτοικοι διαμένοντες στην Νορβηγία. Και καταλαβαίνετε ότι μιλάμε εδώ πέρα για μια πολύ σημαντική νομική ε, αντίφαση. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν δύο πιθανές λύσεις. Πρώτον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Νορβηγία δεν βρίσκεται κάπου στη Λατινική Αμερική ή στην Αφρική. Η Νορβηγία είναι μια χώρα που δύο φορές είπε όχι στην προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Νορβηγία έχει θεσμικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, όταν έχουμε ένα θεσμοθετημένο διάλογο με την Νορβηγία, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα. Το ζήτημα αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τους Ισπανούς εργαζομένους οι οποίοι κατέβαλαν εισφορές στον νορβηγικό προπολογισμό, αλλά έχει να κάνει και με όλους τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι εργάζονταν στα πλαίσια μιας εργασιακής σύμβασης ε, στην Νορβηγία και που κατέβαλαν και αυτοί με τη σειρά τους φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλειας στην Νορβηγία και οι οποίοι τώρα έχουν συνταξιδοτικά δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να λάβουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να θέσουμε το ζήτημα αυτό προκειμένου να λυθεί όχι μόνο η συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και όλες οι άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Δεύτερον, έχουμε και το μέσο των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ισπανίας και της Νορβηγίας. Στην περίπτωση όμως αυτή, αν δεν υπάρχει ευρωπαϊκή διάσταση, μπορώ να φανταστώ ότι η Νορβηγία πολύ εύκολα θα πει «Κοιτάξτε, συγγνώμη, η α, ε, κοινοτική νομοθεσία δεν μας ε, υποχρεώνει να κάνουμε κάτι». Κι όμως υποχρεώνονται γιατί α, ε, θα πρέπει αυτή τη στιγμή δέχονται τα χρήματα και τους φόρους και τις φορές σας από τους Ισπανούς ναυτικούς να τους καταβάλουν και τα συνταξιωτικά τους δικαιώματα. Δεν αναφερόμαστε εδώ πέρα σε παράνομα εργαζομένους, δεν αναφερόμαστε σε μετανάστες, αναφερόμαστε σε συγκεκριμένου πολίτες οι οποίοι έχουν ένα νόμιμο πλέον δικαίωμα και να εργάζονται και να καταβάλουν φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και εν τέλει να λάβουν τα συνταξιωτικά τους δικαιώματα. Καλό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με το ιδιαίτερα ευαίσθητο και σημαντικό αυτό ζήτημα στις σχέσεις που έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση με την Νορβηγία και μια τελική παρατήρηση. Κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται τη κοινωνική δικαιοσύνη, αυτό όντως συγκινεί την αριστερά σκεπτόμενη καρδιά μου, αν θέλετε. Αλλά πρέπει πραγματικά και στην πράξη η κοινωνική δικαιοσύνη να επιτυγχάνεται και στην περίπτωση αυτή των Ισπανών πολιτών οι οποίοι δεν μπορούν να χαίρουν των νομίμων δικαιωμάτων τους. Ευχαριστώ. Όχι, uh, να προσθέσω κι εγώ κάτι. Όντως νομίζω ότι ως Επιτροπή Αναφορών μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με την νορβηγική κυβέρνηση αναφερόμαστε σε μία από τις πιο πλούσιες χώρες στον κόσμο και πραγματικά είναι ντροπή αυτό το οποίο συμβαίνει. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει απλώς να μιλάμε θεωρητικά, αλλά θα πρέπει πραγματικά να επιμείνουμε και να έρθουμε σε επαφή με την νορβηγική κυβέρνηση. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά την χώρα αυτή, συμμετείχα και στο Νορβηγικό Συμβούλιο και πραγματικά νιώθω ότι είναι η δικιά μου η χώρα ουσιαστικά, σαν είναι η πατρίδα μου η οποία συμπεριφέρεται με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να επιληθεί το πρόβλημα αυτό. Μπορεί να μην θέλετε να είστε μέλος Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ ωραία. Αλλά το ζήτημα αυτό υφίσταται και αυτό το οποίο ζητάμε είναι αν μη τι άλλο να είστε ένας εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης τίμιος, ειλικρινής. Νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να θέσουμε το πρόβλημα αυτό και πραγματικά ντρέπομαι εξ ονόματος Νορβηγίας. Οι ε, Ευχαριστώ. Θέλουν οι αναφέροντε να απαντήσουν. Όχι. Ωραία. σα ευχαριστώ όλου ε, για τη συνεισφορά σα. Ε, πρόκειται για μια συνήθιστη περίπτωση. Η ΜΕΝ Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά η ίδια είναι αναρμόδια. Θεωρώ ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, το έχουν ζητήσει άλλωστε όλοι, και δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδρανείς. Ε, θα πρέπει τουλάχιστον να αποστείλουμε μια επιστολή στην ευρυγία και να πιέσουμε περαιτέρω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να ενεργοποιήσει πραγματικά όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να επιταχύνει τη διαδικασία μιας ε, ε, δυνητικής διμερούς συμφωνίας ώστε να πάυσει να υπάρχει αυτή η αδικία όπως αναγνωρίζουν όλοι. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και τους αναφέροντες. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη ή μάλλον τα, επόμενα, διότι έχουμε πάρα πολλές αναφορές. Δεν θα τις αναφέρω μία προς μία. Αναφέρονται όλοι ε, στο θέμα της ε, παράκτειας νομοθεσίας της Ισπανίας. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, θα δώσω τώρα το λόγο στους αναφέροντες. Ε, έχουμε καθορισμένο αριθμό. Εξ ονόματος της Βαλένθια καταρχάς, ο κύριος Χωσέ Ορτέγα, ο οποίος θα μιλήσει από κοινού με την Κάρμεν Τελάνο. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Χωσέ Ορτέγα λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους ε, κυρίους Ευρωβουλευτές. Ε, πολύ γρήγορα. Από την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ δεν έχει αλλάξει και τίποτα σχεδόν. Πράγματι υπάρχει νέο Γενικό Διευθυντή ε, Ακτών, ο οποίος μας έδωσε κάποιες ελπίδες, αλλά να δούμε αν θα υλοποιηθούν. Υπάρχει μια μεταρρύθμιση του νόμου για τις ακτές και εγώ συμμετείχα στην ε, αναδιατύπωση του νόμου αυτούς, αλλά η σημαντική μεταρρύθμιση εξακολουθεί να εκρεμεί και όλα είναι τα ίδια παρά το γεγονό ότι παρενέβη το Κοινοβούλιο. Πέρσι εγώ σα είπα ότι στη Φλωρεντίνα Μαρ της ε, στέρισαν την κατοικία του στη Μαγιόρκα και εξακολουθεί να μην έχει κατοικία. Το πρόβλημα είναι πάντα το ίδιο και είναι ότι εξακολουθεί να ισχύει στην Ισπανία σε αυτή την τόσο φρικτή στιγμή ε, και τα προβλήματα που βιώνει ο Ισπανός ε, ε πολίτης ε, θεωρείται βάσει της Ισπανικής κυβέρνησης ε, άνθρωπος χωρίς δικαιώματα, θεωρείται κλέφτης και αντί να του ζητήσει συγγνώμη του καταδαφίζει την κατοικία του και του ζητά να αποζημιώσει και το κόστος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν υπάρχει αρμοδιότητα για να μελετήσει το θέμα. Στις 20 Ιανουαρίου του 2009 ένας Βρετανός Ευρωβουλευτής είπε στην κυβέρνηση της Βαλένθια «Ακούστε, εσείς δεν ε, προσφύγατε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί έρχεστε εδώ και αναφέρεστε σε κανόνες και νομοθεσία όταν το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι αυτό. Το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να επιλύει τα προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών. Επιτρέψτε μου λοιπόν να συμμεριστώ την άποψή του πλήρως. Μπορώ να συνεχίσω ή πρέπει να ολοκληρώσω. Έχει λήξει ο χρόνος σας γιατί θα πρέπει να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Κάρμεν Τελάμου. Εδώ είμαι. Καλημέρα σας. μισή λεπτό δεν είναι σχεδόν καθόλου χρόνος, επομένως τέσσερα-πέντε πράγματα θέλω να σας πω μόνο και εγώ συμμετείχα στην τροποποίηση της νομοθεσίας, παρόλα αυτά δεν με ικανοποιεί η τροποποίηση της νομοθεσίας που κατατέθηκε και ελπίζω να γίνει σεβαστή η ιδιωτική κατοικία και να επιστραφούν αυτά τα οποία ε, κατασχέθηκαν. Ο παρόν νόμος αποτελεί κατάφορη παραβίαση και αφορά τα δικαιώματα ε, σχεδόν 14 εκατομμυρίων Ισπανών. 14 εκατομμύρια Ισπανών θα υπάρξουν πονοκέφαλοι για πάρα πολλούς Ισπανούς και αυτό σημαίνει ότι θα δώσει δουλειά μεν σε μεγάλες γενναίες ε, δικηγόρων. Αυτοί πραγματικά θα κερδίσουν πάρα πολλά χρήματα, αλλά πρόκειται για ένα ε, νόμο ο οποίος αφήνει ανυπεράσπιστους τους Ισπανούς πολίτες. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι... Ε, είναι καταχραστές ε, δημόσιας περιουσίας ε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Πρόκειται για ένα ε, νόμο ο οποίος είναι κατά του κράτους δικαίου. Αυτές τις φράσεις δεν τις είπα εγώ, τις είπε κανένας εξ ομών. Αυτά αναφέρθηκαν στο Κοινοβούλιο της Ισπανίας όταν συζητήθηκε ο νόμος των ακτών. Θα ήθελα να σας ζητήσω να διαβάσετε αυτές τις μέρες οτιδήποτε αναφέρεται για τον νόμο για τις ακτές. Όλα όσα μπορούμε να πούμε για τον νόμο τις ακτές είναι σε αυτές τις φράσεις. Αυτά είναι λόγια ε, Ισπανών βουλευτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η Μαργαρίτα Γκαρθία Χάιμε τώρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που μας επιτρέπετε να σας απευθύνουμε το λόγο η περίπτωσή μου είναι ανάλογη των ε, σχεδόν 400.000 περιπτώσεων που έχουμε στην Ισπανία, παρά το γεγονός ότι τις αρνείται η Ισπανική κυβέρνηση αυτές τις περιπτώσεις. Θα ήθελα να πω ότι όπως όλοι οι υπόλοιποι είχα μία νόμιμη κατοικία και κινδυνεύω να τη χάσω απολύτως. Το όνομά μου είναι ήδη στον κατάλογο και μου διαβιβάστηκε ότι θα κατεδαφιστεί το σπίτι μου. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι αισθάνομαι ότι με καταδιώκει η κυβέρνησή μου και χρησιμοποιείται ένας νόμος για να με καταλυστεύσουν. Νιώθω ότι είναι ληστρική αυτή η συμπεριφορά και πρόκειται για μια κυβέρνηση η οποία δεν επιτρέπει να συζητηθεί το ζήτημα. Η κυβέρνηση αυτή όχι μόνο μας καταλυστεύει, αλλά αρνείται και ότι συμβαίνει τίποτα στην Επιτροπή Αναφορών. Στην επιστολή που απέστειλε στην Επιτροπή Αναφορών η κυβέρνηση της Ισπανίας, η υπουργό απαντά με ψεύδι. Δεν ξέρω αν απαντά ε, έτσι από άγνοια ή το κάνει εσκεμένα. Αλλά όταν αναφέρεται σε περιπτώσεις που υποστηρίζουν τον νόμο της, αναφέρεται σε περιπτώσεις του Δικαστορίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, της, του Στρασβούργου, που ε, αποφάνθηκαν υπέρ της γαλλικής κυβέρνησης. Τι σύμπτωση όμως, ε, σε αυτή την περίπτωση δεν αναφερόμασταν στην ιδιωτική ιδιοκτησία και ε, μάλλον φαίνεται ότι ο υπουργό είτε δεν ήξερε γιατί μιλούσε ή ήξερε πάρα πολύ καλά σε τι αναφερόταν. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο έχει εκδώσει αποφάσεις που είναι υπέρ των αναφερόντων με πανομοιότυπες περιπτώσεις ε, για την κυβέρνηση της Τουρκίας πανομοιότυπες με το νόμο για τις ακτές της Ισπανίας. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφασίζει κατά της τουρκικής κυβέρνησης αυτές τις περιπτώσεις. Το μόνο λοιπόν που μένει να σας πω είναι ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία που έχει κάποιος και που αγόρασε και δεν έχει καμία σημασία πόσα χρόνια του ανήκε, είναι κάτι το οποίο χάνεται αυτή τη στιγμή ε, χάνουμε το σπίτι μας, ελπίζουμε να ζήσουμε και να πεθάνουμε εκεί και ξαφνικά μας λένε ότι θα μας το πάρουν γιατί υπάρχει ένας νέος νόμος και εγώ θα πρέπει επίσης να πληρώσω για να παλωτριωθεί το σπίτι μου. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή την περίπτωση. Κάποιος θα πρέπει να σκεφτεί και εμάς διότι η Ισπανική κυβέρνηση δεν μας σκέφτηκε ή εάν ε, ε, μας σκέφτεται, μας σκέφτεται με κακόβουλο τρόπο. Πίσω λοιπόν από αυτά τα σχέδια υπάρχουν χωροταξικά σχέδια και όλα έχουν ως κίνητρο ένα ε, μελλοντικό σχέδιο το οποίο ε, θα αποφέρει πάρα πολλά χρήματα και μεγάλες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Χωσέ Ανδρέας Ρουίστελ Μολίνο έχει και μια παρουσίαση PowerPoint η οποία ελπίζω να μην διαρκέσει πάνω από τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι σε τρία λεπτά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας εξηγήσω την έρευνα που έχω κάνει τα τελευταία πέντε χρόνια. Πρόκειται για μία πολύ διεξοδική έρευνα και τα αποτελέσματα ε, δεν μπορούν να φανούν σε μία παρουσίαση PowerPoint. Δεν θα την αναφέρω όλη την παρουσίαση φυσικά γιατί δεν υπάρχει χρόνος ήθελα να δείξω ότι και εγώ και πολλοί άλλοι που ήρθαμε χιλιάδες χιλιόμετρα στις Βρυξέλλες και ξοδέψαμε τόσα ε, χρήματα ε, να έρθουμε εδώ και μας λέτε ότι τρία λεπτά μας δίνετε για πέντε χρόνια κόπο για να τηρηθεί ο περιβαλλοντικός νόμος, γιατί ο νόμος για τις ακτές δεν είναι περιβαλλοντικός νόμος, θα πρέπει να υπάρχουν τρεις συνένοχοι. Η κυβέρνηση της Ισπανίας, η λιμενική αρχή, η παράκτη αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν υψηλά ιστάμενοι της χώρας, ακόμα και μία διευθύντρια της Επιτροπής Παράκτιων ε, Νόμων και η Ισπανική κυβέρνηση δεν ήταν παρούσα εδώ ε, το Μάρτιο για να συζητήσει το θέμα. Παραβιάζεται με τον νόμο αυτό η αρχή της πρόληψης, της προληπτικής δράσης και της ε, διόρθωσης ε, των περιβαλλοντικών σφαλμάτων στην πηγή τους στο άρθρο 8 και 192.2 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται η περιβαλλοντική πολιτική η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νόμος για τις ακτές δεν τηρεί την περιβαλλοντική νομοθεσία. Εδώ έχουμε το λιμένα της Βαλένθια και όλη την περιοχή της Αλμπουφέρα που συμμετέχει στο δίκτυο Natura 2000. Εδώ στην εικόνα αυτή έχουμε την επιδείνωση των ακτών στα νότια του λιμένα της Βαλένθια αυτό προέκυψε βάσει και των μελετών της ε, περιβαλλοντικού αντικτύπου ε, σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος τον Αύγουστο του 2007. Εκεί λέγεται ότι η Ισπανική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για την επιδείνωση των ακτών και θα πρέπει να βελτιωθούν οι ε, συνθήκες εκεί. Και αυτές είναι οι συνέπειες. Τέθηκε σε εφαρμογή οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη τον Οκτώβριο του 2007. Εκεί υπήρχε παραλία, τώρα δεν υπάρχει πια παραλία. Ο Ριπένον δεν πληρώνει. Και όπως σας είπα αυτό δεν συνάδει με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και επιπλέον χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε τι συνέβη. Υπάρχουν τα προγράμματα Life, Ecolite. Ε, εδώ στα δεξιά έχουμε μια περιοχή που είναι στο δίκτυο Natura 2000 ε, και εδώ έχουμε ε, συλλογή της ΣΑΜΟΥ και βλέπετε πού πήγανε όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Swimming in Mediterranean Sea. Εγώ νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να κολυμπήσει σε αυτή τη Μεσόγειο θάλασσα. Και αυτές είναι οι συνέπειες της χρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλο παράδειγμα. η πλειονότητα των Ισπανικών αρχών δεν απάντησαν καν. Εκατοντάδες απεστολές ε, ε, στάλησαν στις Ισπανικές αρχές, κανείς δεν μας απάντησε. Επιπλέον, η κυρία ε, Μουνίδη Τεουρκίσα που είναι εδώ παρούσα, της έχω στείλει τόσα mail και δεν μου απάντησε τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο νόμος για τις ακτές η αρχή Αιγιαλού μας λέει ότι ο νόμος για τις ακτές ε, μας λέει ότι δεν παραβιάζει κανένα δικαίωμα. Επίσης μας λέει, θα περάσω πολύ γρήγορα τις φωτογραφίες γιατί δεν νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να μάθετε την αλήθεια σε τρία λεπτά. Θα τη μάθετε. Θα ήθελα να ξεκινήσει μια έρευνα την Επιτροπή Αναφορών. Πρέπει να κλείσετε σε λίγα δευτερόλεπτα. Σας παρακαλώ λοιπόν να ξεκινήσει μια έρευνα, να μιλήσετε με τους ανθρώπους εγώ είμαι στη διάθεσή σας για συνεργασία, ε, για να δώσω όλη την τεκμηρίωση που έχω στη διάθεσή μου σε αυτή την επιτροπή που θα κάνει την έρευνα. Ο νόμος για τις ακτές παραβιάζει την νομοθεσία και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Τροποποιούν την ε, ε, παράκτια γραμμή και πρέπει εμείς να πληρώσουμε τις συνέπειες και δεν υπάρχει καμία περιβαλλοντική ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ να μην ε, κάνουμε φασαρία εδώ. Θα ήθελα απλώς να διευκρινίσω ότι καθορίσαμε αυτά τα ε, χρονικά περιφέρεια για να μπορέσουν να απαντήσουν όλοι και να υπάρχει και μεγαλύτερη δημοκρατία και συμμετοχή σε αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν είστε ικανοποιημένοι, αλλά η Επιτροπή ασχολείται με το θέμα αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα έχουμε ακούσει. Είναι ευφυές να παρέμβετε σε τρία λεπτά και να μας πείτε τι συνέβη, τι νέο υπάρχει και κάποιο επιπλέον στοιχείο που θα μπορούσε να χρησιμεύσει στην Επιτροπή μας για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και εμείς και να, ε, να αναλάβουμε δράση για να λυθεί το θέμα, το θέμα σας. Χουάνι Τουριμπάρια. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είμαι ιδιοκτήτης μιας κατοικίας που θα γκρεμιστεί. Έχει ήδη γίνει κατάσχεση και παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματά μου. Καταρχήν υπάρχει εδώ μια αναδρομική ισχύ. Βλέπετε τους τίτλους ιδιοκτησίας που έχω από το 1983. Βλέπετε το μητρό, βλέπετε τα αποδεικτικά στοιχεία ότι πραγματικά αυτός ο μήλος μου ανήκει. Πρόκειται λοιπόν για κάτι που δεν μπορεί εδώ να έχει αναδρομική ισχύ. Πρόκειται για μια αυθαίρετη απόφαση. Οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν σε άλλες περιπτώσεις παρόμοιες διατάξεις, φτάνουν σε αντίθετο αποτέλεσμα και παίρνουν διαφορετικές αποστάσεις. Κοιτάξτε που βρίσκεται ο μήλος μου, 7 χιλιόμετρα από την ακτή του Αιγιαλού σε μία περιοχή όπου είναι αδύνατον να γίνει οποιοδήποτε άλλο χορταϊκό σύστημα. Πώς γίνεται λοιπόν η κατάσχετη Παραβιάζεται εδώ η αρχή της νομοθεσίας η οποία ισχύει βάσει μιας μελέτης που έχει γίνει δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτό ο δικαστής ζήτησε μια νέα μελέτη η οποία δεν ελήφθη υπόψη από το δικαστήριο. Το ανώτατο δικαστήριο απεφάνθη βάσει της επιχειρηματολογίας της άμυνας και έφτασε σε ένα αντίθετο αποτέλεσμα. Τι μπορεί κανείς να πει. Έγινε κατάσχεση, δεν είμαι πλέον ιδιοκτήτης αυτής της ε, κατοικίας αυτού του μήλου και διαβάζω εδώ ότι δεν έχω πλέον δικαιώματα, κυρίες και κύριοι, ο νόμος ε, για τις ακτές δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα ιδιοκτησίας. Αν διαβάσει κανείς βέβαια στο άρθρο του αντίστοιχου νόμου, διαπιστώνει ότι υπάρχει αναδρομική ισχύς. Διαβάζω επίσης όσον αφορά τους τίτλους ιδιοκτησίας ότι δεν αναγνωρίζονται τα δικαιώματα αυτά. Εδώ λοιπόν υπάρχει έλλειψη ασφάλειας του νόμου. Πρόκειται πραγματικά για ένα νόμο με αναδρομική ισχύ που παραβιάζει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Τι λέει όμως η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρώπης, κανείς δεν μπορεί να σε καμία περίπτωση μπορεί να παραβιαστεί το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Γι' αυτό και έχω προσφύγει και στο δικαστήριο του Στρασβούργου, αλλά και έχω κάνει και έφεση στην Ισπανία. Παραβιάζονται εδώ τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα δικαιώματα του ανθρώπου και θεωρώ ότι η κυβέρνηση της Ισπανίας θα πρέπει να αναγνωρίσει το θεμελιώδες αυτό δικαίωμα. Sí, sí, sí, estoy aquí. Εδώ πέρα είμαι. Καλημέρα σας. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Ματσόνη και όλους τους ευρωβουλευτές που μας δώσαν τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις του Ισπανικού νόμου περιακτών για όλους τους πολίτες και ιδίω για τους ηλικιωμένους. Έχουμε μια παραβίαση ουσιαστικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν ε, γίνεται σεβαστείο επίσης το τεκμήριο της αθωότητας. Καταγγέλουμε σε κάθε περίπτωση το ότι, μας, ε, το ότι έχουν κατεδαφιστεί πάρα πολλά κτίρια, οι κατοικίες μας, και ουσιαστικά εδώ πέρα θα ήθελα να υπερασπιστώ τους γείτονέ μου, οι οποίοι δεν μιλούν Ισπανικά και οι οποίοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Για αυτούς η κατάσταση είναι χαοτική και δεν μπορούν καν να υπεραμεινθούν των κατοικιών τους, εφόσον δεν μιλούν την Ισπανική γλώσσα. Ένα 98% των περιπτώσεων που κατέληξαν στο δικαστήριο αντιμετωπίζουν την ίδια μοίρα με εμάς. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους και κυρίως ηλικιωμένους που έχουν κατοικίες κοντά στην ακτή. Ενδεχομένως να μην ζήσουμε προκειμένου να δούμε πραγματικά την απόφαση του δικαστηρίου. Δεν θα είμαστε εν ζωή πλέον για να δούμε τι θα γίνει με τις κατοικίες μας και τι απόφαση θα πάρουν τα δικαστήρια. Έχουμε δώσει πάρα πολλά αποδεικτικά στοιχεία, πάρα πολλέ τεκμηριωμένε πληροφορίε για να αποδείξουμε πώ έχει κατάσταση. Πώ μπορεί να λέει τώρα η Ισπανική κυβέρνηση ότι υπάρχει νομική ασφάλεια τη στιγμή που πέρασαν πάνω από 18 μήνες προτού απαντήσουν καν στη δική μας την αφορά, χωρίς να έχουν λάβει καμία δράση ενδιάμεσα. Έχουμε το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναφέρεται στα δικαιώματα στην εξωπρεπή ζωή των ηλικιωμένων. Πρέπει λοιπόν να τροποποιηθεί ο απέσιος αυτός ισπανικός νόμος περιακτών, Πρέπει άμεσα να γίνει κάτι. Θα πρέπει να αναλυφθεί δράση προκειμένου να διορθώσει την κατάσταση της κυβέρνηση. Χωσέ Περές Scusi, stiamo aspettando. Περιμένουμε να μιλήσετε. Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Σας έδωσα το λόγο, παρακαλώ. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Ε, good morning. Ε, I would like to present the case of the shopping center Anexo, Anexo those in Θα ήθελα να αφαιρθώ στο εμπορικό αυτό κέντρο στις Κανάριες ε, νήσους. Πάρα πολλά άτομα εργάζονται εκεί, 6 εκατομμύρια άτομα περνάνε από αυτό το εμπορικό κέντρο, παρέχουμε εμεί πάρα πολλές υπηρεσίες στους ανθρώπους αυτούς. Το 1979 ολοκληρώθηκε το εμπορικό αυτό κέντρο, προτού δηλαδή εγκριθεί ο νόμος αυτός και μάλιστα ακολουθήσαμε ε, την Ισπανική νομοθεσία, καθώς επίσης και τα όσα λέει η κεντρική κυβέρνηση περί ενέγερσης κτηρίων. Το 1958 άρχισαν να μπαίνουν τα πρώτα θεμέλια. Στη συνέχεια, μετά τον νόμο περιακτών του 1969, συνεχίσαμε την κατασκευή και στη συνέχεια βλέπετε πόσο ο επόμενος νόμος, τον οποίο συστάμε αυτή τη στιγμή, άρχισε να καλύπτει και το δικό μας το εμπορικό κέντρο. Βλέπετε λοιπόν πώ λειτουργούν τα πράγματα στην Ισπανία. Αν δεν σα επηρεάσει ο πρώτο ή ο δεύτερο νόμο, δεν την έχετε γλιτώσει. Θα έρθει ένα τρίτο νόμο και θα σα επηρεάσει. Και δεν ξέρουμε αν θα έρθει και ένα τέταρτο νόμο στη συνέχεια. Το 1988 στην τότε νομοθεσία υπόθηκε ότι κάποια κατασκευαστικά υλικά, όπως ακόμα και η άμμος, ανήκουν ουσιαστικά στο κράτος και Κατά αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνετε πώς το ίδιο το εμπορικό κέντρο ε, πέρασε περισσότερο στην ε, δικαιοδοσία του ε, Ισπανικού κράτους. Προσπαθούμε εμεί να δείξουμε, και το έχουμε δείξει και πάρα πολλές αυτές στο παρελθόν, ότι το εμπορικό μας κέντρο συμπεριλήφθηκε, ενώ υπήρχαν άλλα κτίρια, όπως ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο, το οποίο δεν συμπεριλήφθηκε στον, στη δικαιοδοσία του νόμου αυτού. Βλέπετε ότι υπάρχει μια αυθαίρετη εφαρμογή τελικά της νομοθεσίας αυτής. Άρχισε επίσης να ισχύει αναδρομικά, ισχύει όπως σας είπα αυθαίρετα. Εμείς παρόλα αυτά κατασκευάσαμε το εμπορικό αυτό κέντρο εντελώς νόμιμα, ακολουθώντας όλη την νομοθεσία περί αδειοδότησης και περί ανάγερσης κτηρίων, προτού αρχίσει να εφαρμόζεται ο επίμαχος αυτός νόμος. Εμείς καταδείξαμε σε κάθε περίπτωση ότι η νομοθεσία η οποία επιβλήθηκε αργότερα με την ανέγερση του δικού μας του κτηρίου εφαρμόζεται αυθαίρετα. Δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση, προχώρησαν μάλιστα οι Ισπανικές αρχές σε κατάσχεση του εμπορικού αυτού κέντρου. Πιστεύουμε λοιπόν ότι παραβιάζεται το άρθρο 70 της Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς επίσης και διατάξεις ε, της ε, Συνθήκης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και άρθρα της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θεωρούμε λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει κάτι εναντίον αυτού του άδικου νόμου. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου και εμένα να σας κάνω μια παρουσίαση PowerPoint. Καλημέρα σα. Μπορώ στο μεταξύ, επειδή δεν μα δώσετε το λόγο μέχρι ετοιμάζετε την ε, ε, παρουσίαση, να μιλήσω εγώ. Είστε η τελευταία μας ελπίδα. Μα καλέσατε για σήμερα, η πρόεδρο διακόπτη. Όχι, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορεί. Είπα να εκμεταλλευτώ το χρόνο που μου δίνετε. Περιμένετε όμως, γιατί ούτε πια είστε δεν ξέρω. Εάν υπάρχει χρόνος για την παρουσίαση, θα αναστρέψουμε την ε, σειρά των παρουσιάσεων. Τεχνικά προβλήματα. Ενώ λοιπόν βλέπουμε τι γίνεται από τεχνικής πλευράς, θα περάσουμε στην επόμενη. Καλημέρα σας. Μιλήσαμε για την αυτερεσία, για την αναδρομική ισχύ, είπαμε πολλά πράγματα για τον νόμο για τις εχθείς. Ε, η πρόεδρος διακόπτη. Σας παρακαλώ. Θέλουμε πραγματική δημοκρατία. Σας παρακαλώ πολύ. Περνάμε τώρα στον Ζαν Λουίσο Μπίν che non Που δεν είναι παρόν. Τόμας Γκονθάλες Δίαθ. Καλημέρα σας. Επανέρχομαι στο Κοινοβούλιο και τι ελπίζουμε να μας βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να εκφράσω την εγγυλική μου, διότι νόμιζα ότι υπήρχε συμμετοχική δημοκρατία για τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαράδεκτο αφού μας κάνετε να διανύσουμε 4.000 χιλιόμετρα με δικά μας έξοδα, ενώ κανονικά θα πρέπει να τα καταβάλλετε εσείς, να μας δίνετε 3 λεπτά να μιλήσουμε, σε άλλους 1,5 λεπτού και σε άλλους να μην αφήνετε κανένα, καθόλου να μιλήσουν. Εδώ πίσω υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει τις κατοικίες τους και δεν τους βοήθησε κανείς για να μπορέσουν να εκφραστούν ελεύθερα σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου πραγματικά πραγματικά θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχική δημοκρατία. Ενώ εγώ πίστευα ότι θα έπρεπε να υπάρχει, παρόλο που δεν υπάρχει πια στη χώρα μου. Εδώ και ένα χρόνο προσπαθώ να εκθέσω την κατάσταση του χωριού ψαράδων του Ιωβήτου που μας αρνούνται και υπάρχει και μια γενική διευθύντρια που έχει καταδικαστεί από το δικαστήριο και εκπροσωπεί την κυβέρνηση και ψεύδεται ασύστολα ενώπιον του Κοινοβουλίου με χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοροϊδεύουμε Ισπανούς πολίτες, τους παίρνουμε τις κατοικίες τους, ε, τους κάνουμε αστέγους και όπως έλεγε και ο προηγούμενος ομιλητής ε, ε, έχουμε και ηλικιωμένου ανθρώπους. Μας βοηθ... πουλάν τα σπίτια μας στην Ισπανία. Πώς είναι δυνατόν όλος ο αιγιαλός της Ισπανίας ε, να, μας, ε, να μην μας ανήκει και να μας κατεδαφίσουν τα σπίτια μας για να κατασκευάζονται στη συνέχεια κατοικίες για όσους καταχρώνται τα χρήματα της κυβέρνησης και για τους πολιτικούς που τους βοηθούνται. Θα πρέπει να υπάρξει μια επιτροπή έρευνας, διερευνητική επιτροπή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως κάνει και σε άλλες περιπτώσεις. Μια διερευνητική αποστολή η οποία θα πρέπει να πάει επιτόπου σε κάθε μία από τις περιοχές που πλήττονται. Για κάποιους εδώ γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα διότι μας αρνούνται τα ανθρώπινα δικαιώματά μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσπίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία τα ζώα και τα φυτά έχουν περισσότερα δικαιώματα από του πολίτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το δικαίωμα στη διδιοκτησία όμω δεν το αναγνωρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι απαράδεκτο να μα δίνετε το λόγο, είναι απαράδεκτο να μα καταδαφίζουν τα σπίτια μα. Εσεί νομίζετε ότι είναι φυσιολογικό εδώ μέσα σε μια βαλίτσα να είναι ιστορία ενό λαού ή η ιστορια ενό ανθρώπου. Είναι απαράδεκτο να είστε κι εσείς πολίτες ισότιμοι μαζί μας. Για μια φορά τουλάχιστον να έρθετε επί τόπου και να μας δείτε. Έρχεστε εσείς, εμείς σας πληρώνουμε και εμείς ερχόμαστε και, μας πληρώ... και πληρώνουμε μόνοι μας. Πηγαίνετε επί τόπου. Υπάρχουν άνθρωποι που τους δώσατε 1,5 λεπτό. Υπάρχουν ένα σωρό δικηγόροι που τον Αύγουστο ε, μας κατελήστευσαν τα σπίτια μας. Ας έχετε τουλάχιστον μια κάποια εδώ μετά που μας θέρισαν τα σπίτια μας, έρχεται το Σοσιαλιστικό Κόμμα και μας ζητά την ψήφα μας. Αν δεν έχουμε σπίτι, πώς είναι δυνατόν να θέλετε να σας ψηφίσουμε δυόμιση χρόνια μετά που έχουμε μείνει χωρίς σπίτια. Ελπίζω να υπάρξει μια διερευνητική επιτροπή και να έρθει κάποιο με τα χρήματα τη Ευρώπη. Διότι μα σκοτώνεται. Μα σκοτώνετε τη ζωή μα, διότι με τα χρήματά μα καταστρέφεται τη ζωή μα και τα σπίτια μα. Ευχαριστώ πολύ.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 Λυπάμαι που υπάρχουν πάντα τέτοιες ε, έντονα συναισθηματικά φορτισμένες αντιδράσεις και λυπάμαι που οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται τα δικαιώματα των άλλων Ευρωπαίων πολιτών. Είναι περιορισμένος ο χρόνος μας και χρόνος που δίνεται σε εσά πρέπει να δίνεται και στους υπόλοιπους πολίτες των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας δίνουμε το λόγο γιατί θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να μιλήσουν αλλά προσπαθούμε με όριμο τρόπο να βρούμε μια ισορροπία. Σας παρακαλώ λοιπόν για το δικό σας το συμφέρον μην επαναλαμβάνετε τα πράγματα τα οποία έχουμε ακούσει και έχετε ήδη γράψει. Αν είμαστε εδώ και ασχολούμαστε ακόμα με το θέμα, είναι γιατί ίσω έχουμε πρόθεση να σα απαντήσουμε και δεν θέλουμε εμεί να κερδοσκοπήσουμε ει βάρο σα. Δυστυχώ, αυτό είναι το τίμημα τη δημοκρατία. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν έρθει από άλλε περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν και αυτοί δικαίωμα να μιλήσουν. Αυτοί που είχαν έρθει πριν από εσά είχαν το ίδιο δικαίωμα. Σα δίνουμε περίπου δύο ώρε από το χρόνο τη Επιτροπή γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντική η δουλειά αυτή αλλά δεν νομίζω ότι μας αξίζει η αντίδρασή σας. Έντονες αντιδράσεις, υψωμένες φωνές και επικρίσεις για τις εργασίες της Επιτροπής. Και σας το λέω για τους συνάδελφους που ασχολούνται με το θέμα αυτό και όχι για την υποφαινόμενη που σας απευθύνει το λόγο. Αν δεν είναι έτοιμη η παρουσίαση, είστε έτοιμοι, ωραία. Επιστρέφουμε στην Καμπρέλια Μάγερς. Καλημέρα σας. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε τη δυνατότητα να σχολιάσω για άλλη μια φορά την κατάσταση στο νησί της Φορμεντέρα και την δική μου την περίπτωση πιο συγκεκριμένα. Θα ήθελα να σας πω ότι διεκδικώ, όπως και οι υπόλοιποι, το δικαίωμα να τροποποιηθεί αυτός ο άδικος νόμος του 1988 και να σας πω τα βασικά σημεία δικίας που υπάρχει στον Αιγιαλό εδώ και την ε, ιστορία που έχουμε. Όταν μιλάμε για δικία, εννοούμε ότι όλες οι μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νησιού δεν έχουν κατεδαφιστεί, ενώ 45 μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν συμπεριληφθεί στο νόμο. Είναι άδικο κατοικίες οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση πέραν των 100 μέτρων και βρίσκονται και σε δημόσια έκταση ε, να μην έχουν κατεδαφιστεί και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν ε, διεκδικήσει το δικαίωμα αυτό ε, λέει ότι θα του εφαρμοστεί η ίδια νομοθεσία με τον γυαλό που εφαρμόζονταν στο παρελθόν. Είναι αδικία να θεωρούνται δημόσια έκταση κατοικίες οι οποίες είναι κατασκευασμένες πάνω από 100 χρόνια και στα 50 μέτρα από την ακτή να κατασκευάζονται ακόμα νέα κτίρια ακόμα και σήμερα. Πρόκειται για έναν άδικο νόμο, ένα νόμο μέσω του οποίου η Ισπανία καθορίζει τι είναι δικά τη, να περιορίσει τι κατοικίε και να μαστερίσει τι κατοικίε μα από τη μια μέρα στην άλλη. Η Ισπανική κυβέρνηση υπερασπίζεται τον εαυτό τη, λέει ότι είναι πολύ λογικό να ισχύσει ο αναδρομικά ο παράκτιο νόμο και αποζημιώνονται οι προηγούμενοι ιδιοκτήτε. Αλλά ποια είναι η αξία τη προσωρινή εκχώρηση σε μια έκταση η οποία δεν έχει ε, τροποποιηθεί. Κόστος μηδέν. Αυτή τη στιγμή η Ισπανική κυβέρνηση έχει δεκάδες χιλιόμετρα ακτών μηδενικής αξίας. Και λέτε ότι κάποιοι μπορούν να χρησιμοποιούν ε, την παλιά τους κατοικία δωρεάν και ε, για 30-50 χρόνια, αλλά αυτό που δεν λέει είναι ότι μπορεί να κάνει και αναδρομική ε, κατάσχεση της περιουσίας και ότι θα πρέπει να πληρώσει κάποιος ε, για την κατεδάφιση και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Δεν υπάρχει τίποτα και αν δεν υπάρχει κάτι μέσα στον Αιγιαλό Ποιος μας λέει ότι δεν θα αλλάξει σε μερικά χρόνια. Υπάρχει κάποιος από τη Μαγιόρκα που το 2003 του έδωσαν ε, μια συγκεκριμένη έκταση και μετά από δύο χρόνια άλλαξε η έκταση αυτή και θεωρείται ότι βρίσκεται η κατοικία του σε δημόσια έκταση. Ορισμένες από αυτές τις κατοικίες είναι ε, κατασκευές από τσιμέντο, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα σε αυτές τις κατοικίε. Δεν είναι μόνο πέτρε, είναι τμήμα τη ιστορίας και των ονείρων των ιδιοκτητών τους. Στην περίπτωσή μου, το ξενοδοχείο της οικογένειας είναι καρπός του κόπου του πατέρα μου. Πρόκειται για μια επιχείρηση την οποία διαχειριζόμαστε πλέον τα παιδιά του και φροντίζουμε τους πελάτες. Οι μικρές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Φορμεντέρα είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις στην πλειονότητά τους. Το να προσπαθήσετε να κάνετε μια νέα χάραξη των ακτών ε, διακυβεύει το μέλλον του νησιού και είναι χωρίς νόημα, διότι θα μείνουν στα χέρια των τεσσάρων μεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και θα χαθεί η ιδιαιτερότητα του νησιού. Και Όλα είναι σε επιχειρήσεις φυσικά. Είναι άδικο να λέμε ότι πρέπει να μεταχειριζόμαστε έτσι τη Φορμεντέρα, διότι αν η Φορμεντέρα είναι έτσι όπως είμαι σήμερα, είναι χάρη στο λαό της που τη φρόντισε. Και εμείς είμαστε 18 χρόνια στη μάχη για να σταματήσει αυτή η αδικία. Α, τώρα λέμε ότι θα γίνει μελέτη αναπερίπτωση της κατάστασης, αλλά ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι το να δοθεί ικανοποιητική λύση σε όλους τους ιδιοκτήτες δεν θα είναι δυνατό. Γι' αυτό ζητάμε η βεβαιότητα να γνωρίζουμε αν το σπίτι μας ή η επιχείρησή μας θα βρεθεί μέσα στην ε, περιοχή που θεωρείται δημόσια εκδικησία. Συγγνώμη, πρέπει να σας διακόψω γιατί τελείως δεν θα μπορέσουν να μιλήσουν οι πόλοι. Ρόιζα Γκάγια Πόσερ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αφαιρθώ στα χιλιάδες των πολιτών που έχουν επηρεαστεί από τον νόμο αυτών των Ισπανικών περιακτών. Τα περισσότερα από τα σπίτια στα οποία αναφέρομαι κατασκευάστηκαν πριν από την έγκριση της ε, επιμαχής νομοθεσίας. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπαν οι Σας καλώ μόνο να επισκεφθείτε την περιοχή, να δείτε τη βιομηχανική ζώνη να δείτε ότι υπάρχουν όντως κάποιες ζώνες προστασίας και συντήρησης του περιβάλλοντος, ότι υπάρχουν όμως πραγματικά και κατοικίες οι οποίες επηρεάζονται πάρα πολύ από αυτή την νομοθεσία. Οι ιδιοκτήτε αυτή τη στιγμή δεν ζητούν αποζημίωση, ζητούν να μπορέσουν να κρατήσουν τα σπίτια τους. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να δείτε πραγματικά τι κάνει το Δηματικό Συμβούλιο στην περιοχή Επιβάλλεται εδώ πέρα μια ζώνη προστασίας στα 20 μέτρα και υπάρχουν πάρα πολλές κατοικίες οι οποίες κατεδαφίζονται. Δείτε λοιπόν πως έχει η βιομηχανική ζώνη, η οποία είναι κοντά στην περιοχή προστασίας του περιβάλλοντος. Νομίζω ότι αυτή είναι ουσιαστικά πολύ το περιβάλλον και όχι κατοικίες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τώρα με τις παρεμβάσεις. Ο κύριος Γαβριλιάδης, που της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα. Ευχαριστώ. Δεν θα προσθέσω τίποτα καινούριο. Στην παρούσα φάση δεν βλέπουμε εδώ να μπορεί να εφαρμοστεί το κοινοτικό δίκαιο. Παρ' όλα αυτά είμαστε σε επαφή με τις ε, ισπανικές αρχές έτσι ώστε να καθοριστεί αν υπάρχει διακριτική μεταχείριση μη Ισπανών στην περιοχή. Προς το παρόν δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο, δεν έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Συνεχίζουμε πάντως να είμαστε σε στενή επαφή με τις Ισπανικές αρχές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση. Ο κύριος Ιτουργκάιθ, καταρχάς. Ένα λεπτό. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ένα λεπτό μου είπατε ότι έχω. Δυστυχώς, ε, ακόμα και σήμερα, μετά από όσα ακούσαμε, φαίνεται ότι δεν έχει γίνει καμία πρόοδος και η κατάσταση εξακολουθεί να είναι η ίδια. Ακούσαμε και τον αναφέροντα τον ε, κύριο Μπαρία για το μήλο του και το τι συμβαίνει. Εγώ το έλεγα συνεχώς και συνεχίζω να το επαναλαμβάνω. Χρειαζόμαστε ένα νόμο, αλλά ένα νόμο ο οποίος θα είναι συνεκτικός και λογικός. Και εκεί έγινε και το πρόβλημα. Εμείς συνεχώς λέμε και επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε κατά του συγκεκριμένου νόμου, διότι δεν μπορεί να εφαρμόζεται αναδρομικά αυτός ο νόμος. Είμαστε κατά της αυθαίρετης εφαρμογής του νόμου αυτού και θεωρούμε ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή η νομική αβεβαιότητα που δημιουργεί η εφαρμοστική αυτού του νόμου για πολλούς από τους αναφέροντες. Γίνονται κάποια πράγματα στη Γερουσία, το γνωρίζετε, γίνονται πράγματα και στην Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά ο καθένας εκπροσωπεί μια πολιτική ομάδα, ο καθένας έχει ένα διαφορετικό όραμα και διαφορετική πολιτική άποψη για το θέμα αυτό. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι όπως ακούσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δυστυχώς πολύ λίγα μπορούν να γίνουν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς όμως στο πρόγραμμά μας, ε, εγώ το υποστηρίζω, το διεκδικώ και ζητώ από την πολιτική μου ομάδα να διαγραφούν κάποια άρθρα που δεν αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των νομίμων ιδιοκτητών, δεν αναχωρίζουν κάποιες εκχωρήσεις. Πρέπει να σας διακόψω. Διακόπτη Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μέγερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα αυτό επανειλημμένος εδώ στην Επιτροπή μας. Δυστυχώς η Γενική Διεύθυνση Αιγιαλού μας ε, είχε πει ότι θα μας απαντούσε συγκεκριμένα για κάθε μία από τις αναφορές. Δυστυχώς δεν μας έχει διαβιβάσει ακόμα τα στοιχεία και θα πρέπει να αναφέρω δύο, περιπτω... δύο στοιχεία εδώ. Η ομάδα μου συμφωνεί με τον νόμο για τις ακθές. Ο Ισπανικός Αιγιαλός δυστυχώς ήταν ε, ε καταλεηλατημένος και χρειαζόταν αυτός ο παράκτιος νόμος. Δεν συμφωνούμε βέβαια με την αυθαίρετη εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας, διότι πράγματι από το Τσοβίτο στα Κανάρια νησιά μέχρι οποιαδήποτε άλλη περιοχή δεν έχει χρησιμοποιηθεί ένα γενικό κριτήριο και υπάρχει ένα αυθαίρετο κριτήριο το οποίο επέτρεψε να κατασκευαστούν μεγάλες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και ε, δημιουργήθηκε μια πολύ περίεργη κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν έπρεπε να επιλύσουμε το θέμα με πιο αυστηρή ε, εφαρμογή. Κάποιοι όμως ε, ζητάτε να γίνει αυτό διαφορετικά, αλλά θα ήταν σφάλμα δεν μπορείτε να προσβάλλετε όλες τις πολιτικές ομάδες. Είναι σφάλμα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ανδρέασεν. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο νόμος για τις ακτές στην Ισπανία αρχικά είχε καλές προθέσεις. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από την εφαρμογή του νόμου αυτού. Εγώ είμαι Γιού Μαγιόρ και βάσει της νομοθεσίας αυτής υπάρχει μεγάλη νομική ανασφάλεια. Το θέμα της αναδρομικής ισχύω του νόμου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις όπως είδατε και όπως είχαμε ακούσει και την προηγούμενη φορά. Κατάσχεση ιδιωτικής ε, περιουσίας και οι διάφορες κυβερνήσεις προσπάθησαν να επιβάλλουν τον νόμο αυτό δημιουργώντας αυτήν την ασάφεια και ανασφάλεια. Είχαμε υποσχεθεί ένα ειδικό σχέδιο ιδιαίτερα για τα νησιά όπως την ε, Φορμεντέρα. Βλέπετε όμως ότι η αναδρομική εφαρμογή του νόμου αυτού έχει αυξήσει τις ε, δυσκολίες, μικρές οικογενειακές ε, εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, απειλούνται σήμερα και όπως είδαμε υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι επιτόπου υπόσχονται διάφορα τα οποία ποτέ δεν τηρούν. Σήμερα πραγματικά θα πρέπει να σεβαστούμε τα δικαιώματα όλων των Ισπανών, αλλά και όλων αυτών που έχουν έρθει και έχουν εγκατασταθεί σε εμά και σήμερα βρίσκονται σε μια δραματική κατάσταση. Σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πραγματικά θα πρέπει να κάνουμε μια έκκληση στην Ισπανική κυβέρνηση για να κάνει κάτι. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Μούνιτς. Η κυρία. Ευχαριστώ πολύ. Ο νόμος για τις ακτές Υπάρχει από το 1988. Από τότε και με κυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει πολύ. Υιοθετήθηκε παρόλα αυτά δημοκρατικά από το Κοινοβούλιο της Ισπανίας ο νόμος αυτός το 88 και στηρίχθηκε από τις μετέπειτα κυβερνήσεις. Το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο με την απόφαση του 148 του 89 έχει αποφανθεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει άνευ όρων κατάσχεση. Πρόκειται για μια απαλωτρίωση η οποία επιβάλλεται βάσει της νομοθεσίας για τις ακτές ο νόμος αυτός είναι συνταγματικός και πρόκειται για μια δημοκρατική χώρα που δημοκρατικά έχει πάρει τις αποφάσεις αυτής με ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Καταλαβαίνετε ότι και η απόφαση της 29ης ε, Μαρτίου του 2010 στη Γαλλία ε, επιβεβαιώνει αυτή την απόφαση. Ακούσαμε για κάποιες αποφάσεις που αφορούν την Τουρκία. Βλέπουμε όμως ότι η απόφαση στη Γαλλία πάει ακριβώς προς την ίδια κατεύθυνση με τις αποφάσεις των Ισπανικών αρχών. Δεν υπάρχει καμία διακριτική μεταχείριση. Η νομοθεσία αυτή δεν έχει καμία διακριτική επίπτωση και το θέμα είναι η εφαρμογή αυτού του νόμου. Όντως, σε 5% των περιπτώσεων υπάρχουν προβλήματα, 5% των περιπτώσεων ε, διαμαρτύρονται και δεν θέλουν να δεχτούν την εφαρμογή του νόμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο νόμος αυτός περί είναι ένας αναγκαίος νόμος. Είναι ένας περίπλοκος νόμος Όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κοινοτική νομοθεσία δεν έχει παραβιαστεί. Η Ισπανία είναι μια χώρα που βασίζεται στο κράτος δικαίου. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό εδώ. Και θεωρώ ότι υπάρχει γενικότερα μια συνένεση ευρωπαϊκά ως προς αυτό. Υπήρχε μια σειρά καταγγελιών και στο 90% των περιπτώσεων βλέπουμε ότι τα δικαστήρια πήραν μια απόφαση αρνητική για τους προσφεύγοντες. Υποστήριξαν ουσιαστικά την Ισπανική νομοθεσία. Ουσιαστικά εδώ πέρα δεν σας λέω κάτι καινούργιο, επαναλαμβάνω τα όσα έχουμε δει και έχουμε διαβάσει στο παρελθόν. Η δική μας η πολιτική ομάδα είναι προφανώς σε επαφή με τις αρμόδιες εθνικές αρχές και θα προσπαθήσουμε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τους ανθρώπους που πήραν το λόγο. Στην περίπτωση του κύριου Γκαρσία ακούσαμε μάλιστα μια έκκληση η οποία ήταν ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη. Σαφώς εδώ πέρα υπάρχουν πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της αναφοράς και όσον αφορά την χρονική στιγμή κατά την οποία κατατέθηκε η κάθε αναφορά. Αναφερόμαστε πολλές φορές στο συζητήματα όπως η αστική ανάπτυξη, η χωροταξία, Νομίζω όμως ότι η νομοθεσία περί είναι ουσιαστικά μια εθνική νομοθεσία, μια εθνική δικαιοδοσία. Αυτό γνωρίζουν άλλωστε και οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η νομοθεσία αυτή, η οποία υπάρχει ήδη από το 1988, προβλέπει τα όσα ακούσαμε εδώ πέρα. Τροποποιήθηκε βέβαια στη συνέχεια η νομοθεσία αυτή. Και βλέπουμε ότι στην Ισπανία υπήρξε μια πολύ μεγάλη τάση ιδιωτικοποίησης των περιοχών των παράκτιων και αυτό οδήγησε σε πάρα πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα. Σύμφωνα με, την, με το Ισπανικό Σύνταγμα, σαφώς προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι θα πρέπει και η νομοθεσία περί προστασίας των ακτών να συμμορφώνεται με το Ισπανικό Σύνταγμα, όπως ακριβώς θα πρέπει να γίνεται και με την νομοθεσία περί Σαφώς προβλέπεται και η δυνατότητα να προσφύγει κανείς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι είναι δυνατόν να βρεθούν κάποιες γενικά ισχύουσες λύσεις προκειμένου να διορθωθεί η κατάσταση που έχει προκύψει. Ευχαριστώ. Sorry. zwei, drei Punkte. Zum Σας ευχαριστώ. Άκουσα όσοι πήραν το λόγο και προφανώ πιστεύω ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιε λύσει γενικέ υπέρ του γενικού συμφέροντο. Καταλαβαίνετε όμω ότι υπάρχει και η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η οποία ήδη ισχύει εδώ και κάποιο καιρό και η οποία προβλέπει την καταβολή αποζημίωσης περιπτώσει αυτέ. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι πάρα πολλοί αναφέρθηκαν στην αυθαίρετη εφαρμογή τη νομοθεσία αυτή και είπαν ότι πολλέ φορέ το ίδιο το κράτο λειτουργεί ω κλέφτη, ω ληστή τη ατομική περιουσία. Σαφώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία η περίπτωση αυτή, αλλά στην... αν κάναμε κάτι τέτοιο θα ήμασταν απόλυτα άδικοι επένδου στους ανθρώπους αυτούς. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή χάνουν το κεφάλαιό τους, χάνουν την περιουσία τους. Πλήττεται λοιπόν και η ατομική ιδιοκτησία και η ατομική περιουσία, ακόμα και το δικαίωμα μετακίνησης περιουσίας ή αγοράς περιουσίας σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ακόμα και προσβολή του ίδιου του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει εδώ πέρα να βρεθούμε πραγματικά στα δικαιώματα αυτά, καθώς επίσης και στη Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πιστεύω ότι προσβάλλεται στην περίπτωση αυτή η προσυνάρου. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις γιατί αν δεν κάνω λάθος είναι η παλαιότερη υπόθεση αυτή την οποία έχουμε, την οποία συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια χωρίς να καταφέρνουμε να την επιλύσουμε. Πρώτον λοιπόν, επίσημα, καλώ τους αγαπητούς Ισπανούς συναδέλφους να μην παίζουν εδώ πέρα ένα εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι, εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να σας υπενθυμίσω ότι δύο φορές ο κύριος Αφνάρ ήταν στην κυβέρνηση, δηλαδή οχτώ συνολικά χρόνια, και μόνο μετά ήρθε ο κύριος Σταπατέρο. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή οι τελευταίοι να παίζουν τον ρόλο των καλών και να κατηγορούν τους προηγούμενους ότι είναι οι μόνοι κακοί. Σε καμία περίπτωση πάντως εδώ πέρα δεν είμαστε εδώ για να παίξουμε ένα πολιτικό παιχνίδι, για να υποστηρίξουμε το ένα ή το άλλο κόμμα. Πρέπει να δείξουμε στους πολίτες ότι είμαστε εδώ ανεξάρτητα πολιτικών σχηματισμών για να τους υπερασπίσουμε. Είδαμε πολλές φορές ότι οι νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων δεν εντόπισαν παραβίαση της κοινοτική νομοθεσίας. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να αναλάβουν ένα τέτοιο ρόλο προστασίας της εφαρμογής της κοινοτική νομοθεσίας. Δυστυχώς, μάλιστα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας. Προφανώς θα πρέπει να τροποποιηθεί η νομοθεσία αυτή, είναι σαφές. Και δεύτερον, εναπόκειται πλέον στα ισπανικά δικαστήρια να πάρουν μια απόφαση. Και τέλο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί ενδεχομένω και αυτό να αποφασίσει. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννη, παρακαλώ πολύ, σεβαστείτε το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σα. Να νομίζω ότι προσπαθούμε να δούμε την πρόθεση του νόμου, ήταν σίγουρα καλή. Το θέμα είναι όμως ότι δημιουργούνται στην εφαρμογή αυτού του νόμου ε, διάφορα προβλήματα. Βεβαίως το κάθε κράτος έχει δικαίωμα να προστατεύσει τις ακτές του και να χρησιμοποιήσει όλα τα νομικά μέσα για να το κάνει. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι η αναδρομική ισχύ ενός νόμου θα πρέπει να λάβει υπόψη της ε, την ισορροπία μεταξύ των διαφόρων συμφερόντων. Το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των ιδιωτών και να υπάρξουν κάποιες αποζημιώσεις. Ποια είναι τα πλήγματα, αν θέλετε, οι συνέπειες αυτού του νόμου. Ωραία τα σκεφτήκαμε. Υπάρχει και ο νόμος που προβλέπει κάποιες αποζημιώσεις. Το κράτος το δημόσιο συμφέρον προστατεύθηκε. Εδώ όμως βλέπω ότι όσον αφορά τις αποζημιώσεις δεν έχει γίνει αυτό που έπρεπε. Γι' αυτό και θα πρέπει εμείς εδώ να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα αυτών των ιδιωτών που πλήττονται. Είναι απαραίτητο αυτό. Τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας είναι απαραβίαστα και θα πρέπει σαφώς να ληφθούν υπόψη στη γενικότερη αξιολόγηση που γίνεται εδώ. No, no, per favore. Helmer. Uh, thank you, Madam Chairman. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μαρτίνες μας είπε ότι η Ισπανία είναι μια χώρα στην οποία ισχύει το κράτος δικαίου και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Εγώ εδώ το αμφισβητώ. Το αμφισβητώ διότι δεν γίνονται σεβαστά τα ε, δικαιώματα της ε, ιδιοκτησίας που είναι απαραβίαστα και εδώ επιβάλλεται ένας νόμος με αναδρομική ισχύ, κάτι το οποίο είναι αφισβητήσιμο. Θα πρέπει λοιπόν η Ισπανία να δεχτεί αυτήν την κριτική. Η Επιτροπή επίσης είναι εδώ και μας λέει ναι έχουμε διαβουλεύσεις. Εδώ και 10 χρόνια μας λέτε ότι έχετε διαβουλεύσεις και συνεχίζετε να μας λέτε τα ίδια και τα ίδια. Τελικά βλέπουμε ότι η απόφαση της Επιτροπής να μην κάνει τίποτα. Είναι πραγματικά απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Έχουμε γίνει ρεζίλη και σαν Επιτροπή και σαν Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει ρεζίλη, γιατί δείχνουμε ότι μιλάμε για αξίες, για κράτος δικαίου και για δικαιώματα και δεν μπορούμε να προστατεύσουμε ούτε τα θεμελιώδη δικαιώματα για τους κατοίκους της Ευρώπης. Στην ουσία δεν κάνουμε τίποτα. Η κυρία Όκεν. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να αναφερθώ και εγώ σε κάποια πράγματα. Καταρχάς, προφανώς πρέπει να προστατευθεί η ακτή της Ισπανίας. Και αν πραγματικά εφαρμεζόταν σωστά νόμος αυτός από το 1988, εντελώς διαφορετική θα ήταν η εικόνα των Ισπανικών ακτών σήμερα. Δεν μπορεί να είμαστε περήφανοι για αυτήν την εικόνα που έχει η Ισπανική ακτή σήμερα. Βλέπουμε ξενοδοχειακές μονάδες παντού και προφανώς ο νόμος δεν εφαρμόζεται σωστά. Ο τρόπος διαχείρισης νομοθεσίας νομίζω είναι το πρόβλημα, όχι ο νόμος αυτός καθ' αυτός. Τουλάχιστον θα μπορούσαμε να πούμε προς τους πολίτες ότι αν αν έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα από τις τοπικές αρχές, σαφώς θα πρέπει να υποβληθεί κάποια αποζημίωση, αν αποδειχθεί τελικά ότι το λάθος δεν είναι δικός τους. Αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο νόμος αυτός περιακτών διαφέρει από τα υπόλοιπα προβλήματα χωροταξίας που έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να υποβάλουμε μία νέα έκθεση όπου θα ασχολούμαστε μόνο με τον νόμο περιακτών και να αναφέρουμε εκεί πέρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητες. Έχουμε το άρθρο 2 και το άρθρο 7 και μάλιστα μετά τη δική μου την έκθεση ψηφίσαμε για τις αρμοδιότητες αυτές, τις οποίες πλέον επισήμως τις έχουμε και τις οποίες θα πρέπει πραγματικά να προωθήσουμε. Υπάρχουν όντως δικαιώματα εδώ πέρα τα οποία παραβιάζονται. Ευχαριστώ. Κυρία Χιμένες. Ε, ναι. μόλις έμαθα ότι υπάρχουν και κάποιοι Ισπανοί πολίτες από το Κάντιθ, από την περιοχή μου στην Ανδαλουθισία, οι οποίοι δεν θα έχουν χρόνο ομιλία. Γι' αυτό λοιπόν θα χρησιμεύσω εγώ ως ε, φωνή των ε, γεωργών και των ε, κατοίκων της περιοχής του Κάντιθ, διότι είναι οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο ο νόμος για τις ακτές επιτίθεται σε αυτές τις επιχειρήσεις με σημαντικές οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Τους ε, στερούνται οι επιχειρήσεις τους ε, και τους δίνεται μία ελάχιστη αποζημίωση. Η απόφαση του δικαστηρίου έχει δημιουργήσει τεράστια νομική αβεβαιότητα και εμείς έχουμε το καθήκον να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα των νομίμων ιδιοκτητών. Η Ισπανική κυβέρνηση θα πρέπει να διορθώσει αυτές τις παρατυπίες, ε, διότι πρόκειται για ένα νόμο ο οποίος έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για τη ζωή ε, εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών και στην εικόνα της Ισπανίας. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς δεν μπορούμε να τους απογοητεύσουμε, διότι μας κοιτούν στα μάτια, είμαστε η τελευταία τους ελπίδα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τους καταλάβουμε και να τους εισακουστεί η φωνή τους όπου είναι απαραίτητο. Θα ήθελα να πω ότι αυτό που δεν μας αρέσει είναι ότι εδώ γίνεται μια αντιπαράθεση η οποία μας οδηγεί σε ένταση. Δεν μου αρέσει επίσης το ότι αυτή εδώ η η Επιτροπή γίνεται κατά κάποιο τρόπο ο τόπος όπου συνεχίζονται εθνικές αντιπαραθέσεις, διαμάχες και διαφωνίες. Καταλαβαίνουμε ότι η Ισπανική κυβέρνηση έχει κάνει κάποια πράγματα για να προστατεύσει τα δικαιώματα, αλλά όχι αρκετά. Υπάρχει μια νομολογία, η νομολογία η οποία ορίζει ότι όχι απλώς το κοινοτικό δίκαιο θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν πρέπει να προστατευτούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά, αλλά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, στην περίπτωση όπου περιορίζονται, συρρυκνώνονται δικαιώματα των πολιτών. Και σε αυτή την περίπτωση, και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων να υπερισχύσει. Ακούσαμε πραγματικά όλους αυτούς που πήραν το λόγο. Είναι ένα περίπλοκο θέμα και σας παρακαλώ πολύ δώστε μου λίγο παραπάνω από ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Πρέπει να ακουστούν όχι μόνο τα πραγματικά γεγονότα, αλλά θα πρέπει η νομική υπηρεσία να αποφανθεί εδώ. Και θα ήθελα να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Στο ρωμαϊκό δίκαιο υπάρχει η αρχή η οποία εδώ θα πρέπει να είναι απαραβίαστη όσον αφορά τα ισπανικά δικαστήρια στην παρούστα υπόθεση, θα πρέπει να υπάρξει η αναγνώριση της παραβίασης του κοινοτικού δικαίου, κάτι που σημαίνει ότι θα διακοπεί η διαδικασία ενώπιον των Ισπανικών δικαστηρίων και ότι θα υπάρξει προδικαστικό ερώτημα το οποίο θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό σημαίνει ένα συγκεκριμένο χρόνο. Η κυρία Μπιλπά Μπαραντίκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας πω μόνο ότι ίσως ο Ισπανικός νόμος να ήταν απαραίτητος. Δεν λέω όχι, αλλά από τις περιπτώσεις που γνωρίζω και από τις αναφορές που έχουν γίνει στην περιοχή, θεωρώ ότι έχει γίνει μια ακατανόητη διαχείριση των θεμάτων αυτών, όπως έγινε με το μήλο του κυρίου. Και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι καταφεύγουν σε διάφορους οργανισμούς και δαπανούν χρήματα. Ε, θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια σωστή διαχείριση. Και αυτό περιμένουμε να ακούσουμε από τις Ισπανικές αρχές. Όποιος και αν είναι υπεύθυνο να αναλύει την κάθε περίπτωση και να δίνει την κατάλληλη λύση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να βρίσκονται μεσοπέλαγα χωρίς καμία λύση. Δεν υπήρχε καμία διαφάνεια, δεν γνωρίζουμε με ποια κριτήρια καθορίζεται ο γυαλός και θα πρέπει ε, να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βοηθήσουν οι αρμόδιες αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι δεν μπορεί να Ευρωπαϊκής στα θέματα αυτά, διότι δεν υπάρχει διάκριση με την εφαρμογή της νομοθεσίας και είναι κρατική νομοθεσία αυτή. Το ίδιο συμβαίνει και με τον νόμο και άλλους νόμους που διαχειριζόμαστε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν υπάρχει λοιπόν μία απόφαση, πολλοί από τους ευρωβουλευτές και από τις πολιτικές ομάδες αυτό που λένε είναι ότι δεν μπορούμε να επισέλθουμε στα ιστορικά θέματα. Εγώ λοιπόν προτείνω να, επειδή η διαχείριση είναι ακατάλληλη, επειδή δεν υπάρχει καμία διαφάνεια και δεν υπάρχουν κατάλληλες λύσεις, να προσπαθήσουμε από κοινού να λύσουμε το θέμα το. Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω των εκθήσεών μας είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Αλλά χρειαζόμαστε κατεπήγοντα μέτρα και κατεπήγουσες λύσεις για τις διακρίσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Καταρχήν ζητώ συγγνώμη γιατί δεν ήμουν ε, σε όλη την ε, διαδικασία παρούσα. Έπρεπε να ψηφίσω σε μια άλλη επιτροπή. Έχουμε υποβάλει ερώτημα στην αρμόδια επίτροπο, στην κυρία Ρέντινγκ. Και πραγματικά θεωρώ ότι η Επιτροπή θα πρέπει εδώ να αποφανθεί για το κατά πόσον ξένοι, δηλαδή όχι οι Ισπανοί υπήκοοι, πλήττονται από αυτόν τον νόμο. 90% αυτών που έχουν εδώ υποβάλει τις αναφορές δεν είναι Ισπανοί υπήκοοι. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν έχουν γίνει κάποιες έρευνες από μέρους της Επιτροπής για το θέμα αυτό της διακριτικής μεταχείρισης. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουν γίνει καταγγελίες για παραβιάσεις ανάλογες εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Επιτροπή Αναφορών και έχουν επηρεαστεί αρνητικά πάρα πολλοί πολίτες. Πρέπει να σταματήσουμε πλέον να μιλάμε θεωρητικά και να αναλάβουμε πραγματική δράση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να λέει ότι δεν έχουν αρμοδιότητα όσον αφορά το πρόβλημα αυτό. Πρόβλημα που έχει να κάνει με τα δικαιώματα περιουσίας, δικαιώματα ιδιοκτησίας. Και υπάρχουν πολλοί πολίτε που λένε ότι στην περίπτωση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματά του. Αυτό που συμβαίνει όμω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να χρηματοδοτεί τι περιφέρειες αυτέ όπου λαμβάνουν χώρα οι παράτυπε αυτέ διαδικασίε. Και είδαμε εδώ πέρα και κάποια παραδείγματα από τους ίδιους τους αναφέροντες. Για ποιο λόγο λοιπόν εμείς συνεχίζουμε και χρηματοδοτούμε τις περιφερειές αυτές όπου λαμβάνουν χώρα αυτές οι παράτυπες διαδικασίες. Έχω υποβάλει τροπολογίες στον προπολογισμό του 2012, το κοινοτικό, όπου ζητώ να σταματήσει η χρηματοδότηση προς περιφέρειες αυτές, όπου έχουμε δει τα φαινόμενα αυτά και ελπίζω ότι οι συνάδελφοί μου στην αίθουσα αυτή θα στηρίξουν αυτές τις τροπολογίες Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να παρέμβει για να απαντήσει τώρα. Ε, ε, Ευχαριστώ. Ακριβώ αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε με τι ισπανικέ αρχέ. Μιλάτε για 90-95% Πού το βρήκατε αυτό τον αριθμό. Εγώ μέχρι τώρα έχω δει ότι η μεγάλη πλειοψηφία είναι Ισπανοί υπήκοοι, οι οποίοι πλήττονται από τον νόμο αυτό. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν είναι Ισπανοί. Αυτό που το βρηκατε αυτο τον αριθμο εγω μεχρι τωρα εχω δει οτι η μεγαλη πλειοψηφια ειναι ισπανοι υπηκοοι οι οποιοι πληττονται απο τον νομο αυτο αυτο δεν σημαινει βεβαιως οτι δεν υπαρχουν και καποιοι αλλοι οι οποιοι δεν ειναι ισπανοι Από όσο προσπαθουμε να δούμε με τις Ισπανικές αρχές είναι να διερευνήσουμε αν υπάρχει διάκριση για μη Ισπανούς και αυτό προσπαθούμε να διερευνήσουμε και τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ τον ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα. Έχετε ελέγξει αν υπάρχουν τρόποι να Πούμε εδώ ότι υπάρχει θέμα ε, διαγωνισμών και δημόσιων ε, διαδικασιών στην περίπτωση αυτή στην Ισπανία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, αυτό που μας ρώτησε ο συνάδελφος είναι για την περίπτωση εκχώρησης κάποιων ε, έργων ή κάποιων τμήματων της γης στην περιοχή αυτή, το δικαστήριο έχει ήδη αποφανθεί, ακούσαμε τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όσον αφορά τον νόμο για τις δημόσιες προμήθειες δεν εφαρμόζεται εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις. Περιμένουμε βέβαια και την τελική απόφαση και μόλις είναι διαθέσιμη η απόφαση αυτή θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Grazie. Allora, stavo ehm, adesso dando la parola. Ωραία. Έδινα το λόγο για να απαντήσουμε τώρα στους αναφέροντες όπως έχει διαδικασία. Για λόγους οργάνωσης των εργασιών θα δώσω καταρχάς το λόγο σε άλλους ε, τόσους αναφέροντες όσους παρενέβησαν στην αρχή, άλλους δέκα. αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε σε δέκα άλλους αναφέροντες το λόγο και όχι σε αυτούς που ήδη παρενέβησαν. Ξεκινάμε λοιπόν τη διαδικασία απάντησης. Η απάντηση είναι για ένα λεπτό. Σας παρακαλώ τηρήστε τα χρονικά όρια. Χουάν Χιμέρα. Καλημέρα σας. Καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την ε, παρέμβασή μου, αλλά δυστυχώς ε, ε, θεωρούμε ότι η κατάσταση είναι πονίδιστη. Δεν κάνω πολιτική, δεν είμαι υπέρ του ενός ή του άλλου. Τον εαυτό μου υπερασπίζομαι, την οικογένειά μου. Δεν είμαστε μεγάλοι γείτονε, είμαστε μία οικογένεια. Έχουμε ένα σπίτι στα νότια της Μαγιόρκα και η οικογένεια μου εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση στην ίδια περιοχή τα τελευταία 50 χρόνια. Έχουμε περάσει από ηλεκτρική ενέργεια μέσω άνθρακα, έχουμε δηρώσει τον χώρο, ε, φυσικό χώρο ειδικού ενδιαφέροντος, ε, συμμετέχει και στο δίκτυο Natura 2000 και παρόλα αυτά, μετά από όλα αυτά, δύο χρόνια αργότερα έρχεται αυτός ο διάσημος νόμος για τις ακτές και μας ε, ε, κατασχόνται 70 εκτάρια με κατοικίες στην περιοχή. Επαναλαμβάνω, είμαστε μία οικογένεια και είμαστε πλήρως ανυπεράσπιστοι. Θα ήθελα να πω εδώ ότι στην περίπτωσή μας μία έκταση 15 μέτρων λέγεται ότι είναι ε, παραλία και δεν υπάρχει τίποτα γύρω. Δεν είναι αλήθεια. Η παραλία αυτή υπήρχε εδώ και 6.000 χρόνια και εδώ τώρα ένας βούρκος είναι. Εφαρμόζεται ο νόμος για τις ακτές 7.000 χρόνια πίσω στην ε, περίοδο. Πρόκειται για βαρβαρότητα λοιπόν. Οι άνθρωποι που καθόρισαν την ακτή ε, ένα χρόνο αργότερα ε, αφαιρούν ένα σύστημα και εκεί έχουμε 1500 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μόνο μία μικρή έκταση βρίσκεται μέσα στην περιοχή της παραλίας. Μας εκμεταλλεύονται ε, και μας χάνουμε όλη την έκτασή μας. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να σας διακόψω. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα απλώς ε, να πω κάτι. Υπάρχουμε ε, μια εγκεκριμένη εκτογραμμή από το 2003 βάσει του ίδιου νόμου που δεν επηρεάζει καμία από την, ε, καθόλου από την έκτασή μας και τρία χρόνια αργότερα έρχονται και μας παίρνουν την έκτασή μας. Αυτό είναι αυθαιρεσία. Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάρεν Κόμπερλινγκ. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Θέλω να πω κάτι στον κύριο Μαρτίνες, ο είναι τόσο σίγουρος για το κράτος δικαίου. Εδώ και 33 ζω σε ένα μικρό ψαροχώρι στην περιοχή Φαρμοντούρα και πραγματικά αγαπώ αυτήν την περιοχή και είμαι υπήκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζω με τους Ισπανούς στην περιοχή εδώ και χρόνια. Πραγματικά θέλω να σας πω ότι αυτά που συνέβησαν δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που περιγράφονται. Υπήρξε μία πρόταση του Δήμου η οποία τελικά δεν ε, Πρόκειται για ένα φυσικό πάρκο το οποίο έχει αναγνωριστεί και χαρακτηριστεί σαν φυσικό πάρκο και την ίδια ώρα βλέπουμε να υπάρχουν σχέδια χωροταξικά. Είναι προστατευμένη περιοχή και θαλάσσια και χερσαία και την ίδια ώρα βλέπουμε να υπάρχουν σχέδια ανοικοδόμησης. Εγώ ζω εκεί, είμαι καταχωρημένη στα Μητρώα των κατοίκων, πληρώνω φόρους και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι καταπατούνται τα δικαιώματά μου και υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις, παράνομες. Είμαι μία ξένη, αν θέλετε, στην περιοχή και βλέπω τις Ισπανικές αρχές να ανακοινώνουν μια ωραία μέρα ότι πρόκειται για δημόσιο τομέα, δημόσια ιδιοκτησία. Χρειάζομαι λοιπόν κάποια στιγμή να ακουστεί η φωνή μας. Είμαστε διατεθειμένοι να αποδείξουμε αυτά που σας λέμε και είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε οτιδήποτε θέλετε. Είμαστε πραγματικά στη διάθεσή σας, αλλά χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας. Θέλω και τεκμηρίωση. Αν πραγματικά έχετε αποδείξει, σας παρακαλώ να μας τις δώσετε και γραπτός ε, για να τα δώσετε στη γραμματεία και να καθορίσουμε και την απόφασή μας βάσει και τις τεκμηρίωσεις που θα μας δώσετε. Γιάν Φανσούβινσαν τώρα. Ε, Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση αυτή. Όταν φτάσαμε, ενημερωθήκαμε επίσης και για την πορεία την οποία ακολουθεί η αναφορά μας, η οποία υποβλήθηκε το 2010. Λάβαμε επίσης και τις παρατηρήσεις, καθώς επίσης και την απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου γίνονται κάποιες γενικές παρατηρήσεις στο κεφάλαιο 3 καθώς επίσης και μία αναφορά στο κεφάλαιο 4. Ενδιαφέρουσα η απάντηση αυτή. Είδαμε ότι ανελήφθη η δράση και ότι η Ισπανική κυβέρνηση αναγκάστηκε να απαντήσει στο δικό σας το αίτημα. Ωστόσο, δεν είχαμε πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, οι οποίες απεστάλησαν από την Ισπανική κυβέρνηση και η μελέτη αντικτύπου στο περιβάλλον ουσιαστικά αναφέρεται σε αυτό το οποίο εμείς ακριβώς καταγγέλουμε μέσω της αναφοράς μας. Θεωρούμε ότι ε, η νομοθεσία αυτή, και αυτό άλλωστε φαίνεται και στην ε, απάντηση αυτή, δεν εφαρμόζεται με το σωστό ε, τρόπο και έχει βέβαια και την υποστήριξη της κοινοτικής χρηματοδότησης. Πρέπει να πω βέβαια ότι τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντιτάσσονται στα πραγματικά γεγονότα, γιατί αν διαβάσετε την δήλωση της ισπανική κυβέρνησης όσον αφορά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, όπως ακριβώς απορρέπει του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και να συγκρίνεται αυτό με αυτό το οποίο εμεί λέμε συνεχώς, βλέπετε αμέσως ότι τα συμπεράσματα δεν είναι σωστά και ότι ουσιαστικά είναι το αντίθετο από την πραγματική κατάσταση. Λέτε ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι υπήρξε σοβαρή παραβίαση των ε, κοινοτικών οδηγιών κατά την εφαρμογή του σχεδίου αφού το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από τα διορθωτικά ταμεία. Και λέω ότι το σχέδιο αυτό ε, διακόπτη πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Cliff Carter. Θα ήθελα να πω ότι περιμένουμε περαιτέρω δράση από την Επιτροπή Αναφορών. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ωστόσο, μία έκθεση ακόμα ενδεχομένως να βοηθούσε το όλο σύστημα να λειτουργήσει καλύτερα και θα προωθούσε την όλη υπόθεση. Θα μπορούσαμε κατά αυτόν τον τρόπο να διερευνήσουμε ακόμα καλύτερα τα δικαιώματα αυτά ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό αυτή όμως επίπεδο. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η διαδικασία αυτή και σας κάνω αυτή τη στιγμή μια εκκλησία. Ας μην σταματήσουμε τώρα. Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή μέχρι να καταφέρουμε τουλάχιστον να έχουμε μια κάποια αποζημίωση, μια διόρθρωση της κατάστασης. Η νομοθεσία του 1988 άλλαξε τον ορισμό της ε, ιδιοκτησίας, της δημόσιας ιδιοκτησίας και ουσιαστικά πάρα πολλοί ιδιώτες βρέθηκαν να υπόκεινται από τη μία μέρα στην άλλη σε αυτές τις νέες διατάξεις της δημόσιας ιδιοκτησίας. Δεν μπορούμε όμως να αποδεχθούμε ότι το κράτος μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να παίρνει τα σπίτια μας χωρίς να προσφέρει καμία απολύτως αποζημίωση. Διακόπτη πρόεδρος. Δεν θέλουμε όμως εμείς αποζημίωση. Αυτό που θέλουμε είναι τα σπίτια μας. Θέλουμε την ιδιοκτησία μας. Χιμένες Ντομίνκο. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να δώσω κάποια στοιχεία επιπλέον, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ένα χρόνο αργότερα, δυστυχώ, καταγγέλνουμε και πάλι τα ίδια που καταγγείλαμε και την προηγούμενη φορά. Το χρόνο μα χάνουμε και μόνο. Και εμεί και εσεί. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε σεβασμό και εσείς μας αξίζετε και εσείς το σεβασμό στον εαυτό σας. Υπάρχει μία εκμετάλλευση, δεν υπάρχει καμία αποζημίωση χρηματική και πρόκειται για κατάχρηση. Αναδρομική ισχύ στο ρωμαϊκό δίκαιο απαγορεύεται και εδώ υπάρχει και ενοχή. Για παράδειγμα, το εργοστάσιο του 1860 του Φεϊτέρο τώρα κατά πάσα πιθανότητα θα απολωτρωθεί. Στο πλάι, πολύ κοντά, έχει δοθεί έγκριση χρήσης για 40 χρόνια ακόμα της περιοχής ε, ε, του δηληστηρίου του Πετρονό. Ε, όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό μολύνει περισσότερο και ρηπαίνει περισσότερο από την άλλη περιοχή, αλλά έτσι έχουν τα γεγονότα. Και αυτό νομίζω ότι είναι αδικία. Η σύγκριση τώρα της αξιολόγησης περιβαλλοντικού αντικτύπου. Τι μας λέει. Υπάρχει μία αγορά που λειτουργεί. Η διοίκηση γίνεται μέσω επιχειρήσεων, οι οποίες με τη σειρά του δυστυχώ πρέπει να ολοκληρώσετε. Παρουσιάζονται τα σχέδια και οι επιχειρήσεις που εργάζονται μόνο για την ε, διοίκηση δημιουργούν μια κατάσταση που ενώπιον των δικαστηρίων αποδεικνύει πράγματα τα οποία είναι τελώς αντίθετα με αυτά που έχει κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση δημιουργείται ένας μηχανισμός απόλυτης αλήθειας. Και αυτό είναι τρομακτικό. Ραμόν Σόουζα. Καλημέρα σας. Η μητέρα μου είναι ιδιοκτήτρια μιας ιδιοκτησίας που κατασκευάστηκε το 1506 και είναι εγγεγραμμένη στα Μητρό από το 1684. Πλέον δεν της ανήχει το στέρισε ο παράκτιος νόμος του 1988. Η κατάσταση αυτή κατέστρεψε τη ζωή μας, την υγεία μας και την οικονομική μας κατάσταση. Εσείς ήσασταν η τελευταία μας ελπίδα. Μας καλέσατε εδώ και μας είπατε ότι θα εξετάσετε την αναφορά μας. Ζητώ συγγνώμη, αλλά μας ε, διακόψατε, δεν μας επιτρέπετε να μιλήσετε. Εσείς έχετε βάλει έξι αιώνες κληρονομιάς και πάνω από 40 χρόνια ε, προβλημάτων σε 8 γραμμές. Αυτό μπορούμε να πούμε μόνο και δυστυχώς δεν εγκατοπτρίζεται η κατάστασή μας και δεν υπάρχει καμία λύση για τα προβλήματα των Ισπανών και των Ευρωπαίων. Μας έχετε κοροϊδέψει και μας έχετε απογοητεύσει και εμείς αλλά και όλοι όσοι δεν έλαβαν το λόγο είναι απογοητευμένοι. Εσείς μας πήρατε το τελευταίο που μας έμενε, τη φωνή, την ελπίδα και την εμπιστοσύνη στην Επιτροπή Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Αντώνιο Λόνθο. Αντώνιο Λόνθο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος επειδή δεν έχουμε χρόνο. Για μένα ο παράκτιος νόμος δεν με κλέβει, αλλά μου κατέσχεσε πράγματα. Εγώ έχω όλα τα στοιχεία εδώ. Δυόμιση χρόνια. Δυόμιση χρόνια είμαι άστεγος. Και η ισπανική κυβέρνηση, η χώρα μου, γιατί νιώθω ισπανός, δεν γνωρίζω ούτε που μου διαμένω. Υπάρχει μία πράξη από το 1953 η οποία μου στέρισε τη μοναδική μου κατοικία, τα μοναδικά μου επιπλά και τη μοναδική μου ιστορία. Όλα βρίσκονται σε χαρτιά τα οποία δεν υπάρχουν, σε ερήπια τα οποία δεν υπάρχουν. Η κατοικία μου κατασκευάστηκε νομ, νομίμως με τις άδειες του 1953. Έχω και πιστοποιητικό της ασφάλειας της Ισπανίας που μου ε, κάνει πλήρη κατάσχεση και απαλωτρίωση εδώ και δύο χρόνια. Οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές αρχή, ε, της Ισπανίας δεν γνωρίζουν ούτε που διαμένω αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι αυτό το επωνίδιστο κυρίες και κύριοι. Το πιο επωνίδιστο είναι ότι υπάρχουν ε, ανάλογες περιπτώσεις με μένα πάρα πολλές πάμπολες. Στα Κανάρια υπάρχουν παραδοσιακές κατοικίες οι οποίες αντί να διατηρηθούν για να διατηρήσουμε την ποικιλομορφία και την ιδιωτερότητά τους με τα μία τα οποία και κονδύλια τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαφανίζονται βαθμιδών. Υπάρχουν μήλοι, υπάρχουν κατοικίες, υπάρχουν πάρα πάρα πολλές κατοικίες. Και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, διότι ε, μας γίνεται πραγματική αφέμαξη, πηγαίνουμε από δικηγόρο σε δικηγόρο να βρούμε το δίκαιο μας και κανεί δεν μας το δίνει. Ευχαριστώ πολύ. Χουάν Χωσέ Αγκόστο. Καλημέρα σας. Εκπροσωπώ την Τόρε Λασάλ. 50 οικογένειες πλήρωσαν πάνω από 1000 ευρώ για να βρίσκομαι εδώ σήμερα, γι' αυτό σας παρακαλώ αφήστε με να εκμεταλλευτώ αυτό το ένα λεπτό. Το 1957 γίνεται μία χάραξη της ακτογραμμής ε, και υπάρχουν κάποιες κατοικίες οι οποίες θα πρέπει να μείνουν απ' έξω. Ο νόμος όμως ο υπουργικός ο οποίος ε, απαγόρευσε αυτό τον Αιγιαλό είπε ότι δεν ισχύει πλέον η κατάσταση και δημιουργήθηκε νέος Αιγιαλός και επιλέχθηκαν κάποιες ε, κατοικίες οι οποίες έχουν κλειστεί σε ένα πλήρες τετράγωνο. Έχουμε μια νέα χάραξη στη συνέχεια και εγκρίνεται με νέο Υπουργικό Νόμο εκτός από τις κατοικίες αυτές οι οποίες βρίσκονται στην ε, χάραξη του 1957. Εμείς βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα νομικό λίμπο. Δεν ε, εντασσόμαστε ούτε στο 57 ούτε στο 93 τη χάραξη της ακτογραμμής. Αλλά οι αρχές της Ισπανίας ε, ενώ είναι τόσο εύκολο να χαράξουν ε, ένα σχέδιο και δεν τους κοστίζει τίποτα να μας εντάξουν σε κάποιο νόμο. Κάθε φορά που έρχεται κάποιος όμως που θέλει να κάνει κάτι, μας επιβάλλει πρόστιμο. Εσείς μας λέτε να προσφύγουμε στα δικαστήρια. Όταν το συζήτησα εγώ από κάποιον από τη δικαιοσύνη, μου είπε ότι ακόμα και αν προσφύγετε στο δικαστήριο, την επόμενη ημέρα ο παράκτιος νόμος θα χαράξει ένα νέο οικιαλό και δεν θα σας περιλαμβάνει στην, στο σχέδιο πόλης. Ε, οπότε και τι να πάμε να κάνουμε στο δικαστήριο. Σας ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση. Im, im, im von ναι. ναι. Λοιπόν, το 2009 το Μάρτιο η κυρία Όκεν στην έκθεσή της, στο σημείο Π, διαβάζω όσον αφορά την χάραξη της γραμμής, ο σχεδιασμός έγινε καθαρά αφαίρετα και έπληξε κυρίως ξένους κατοίκους της περιοχής. Θα ήθελα εδώ να πω δίνοντάς σας το δικό μου προσωπικό παράδειγμα. Στη δική μας παράκτια περιοχή έχουμε ένα μικρό σπιτάκι, 180 μέτρα από την θάλασσα. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν δύο τεράστια ξενοδοχεία. Το ένα από αυτά ανήκει σε έναν πρώην γερουσιαστή. Θέλω να σας πω ότι η γραμμή αυτή δεν τηρείται σε αυτή την περίπτωση. Τα ξενοδοχεία αυτά απέχουν 20 μέτρα από τον Αιγιαλό. Κύριε Μαρτίνες, ακούστε με και λάβετε γνώση αυτών που σας λέω. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συζήτηση. Είμαι πεπισμένη ότι είναι θετική η πρωτοβουλία μας παρά το γεγονός ότι όπως λέγεται στα μέρη μου όπως και να το κάνεις, ε, λάθος κάνεις. Ε, αντιλαμβάνομαι από τις επικρίσεις ε, προς την Προεδρία ότι θεωρείται ότι είναι λάθος μου που δεν έδωσα το λόγο τους περίπου 100 παρισταμένους και παραπάνω. Ε, Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι ανέλαβα και τήρησα σωστά τη σημερινή μου δέσμευση. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους αναφέροντες που δεν είχαν τη δυνατότητα να παρέμβω, αλλά και όλους αυτούς που παρενέβησαν, αν έχουν υλικό ή τεκμηρίωση που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη στην Επιτροπή μας για να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε, να το παραδώσουν στη Γραμματεία ακόμα και τώρα στη λήξη των εργασιών της Επιτροπής μας. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ περίπλοκη και το θέμα είναι πολύ περίπλοκο και γι' αυτό ακριβώς ε, θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους ε, να αναστείλουμε την απόφαση ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε ε, πιο επισταμένα όλες τις παρεμβάσεις που ακούσαμε και τα έγγραφα τα οποία θα μας παραδοθούν και να λάβουμε απόφαση αργότερα η οποία θα είναι πιο κατάλληλη. Αυτό το οποίο προκύπτει από τη συζήτηση είναι ότι ακόμα και τώρα μετά από τόσο καιρό υπάρχει στέρηση δικαιωμάτων και μία νομοθεσία που ε, παραβιάζεται όπως ακούγεσαμε σε όλες τις παρεμβάσεις. Δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι θα επιρρύψουμε ευθύνες. Ε, Δυστυχώς ε, έτσι έχουν τα πράγματα. Υπάρχουν ε, δικαιώματα τα οποία παραβιάζονται και εμείς έχουμε καθήκον να παρεύουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να μας λέει ότι δεν έχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα από του θέματος και εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να παραβιάσουμε την αρχή της επικουρικότητας σε εθνικά θέματα, αλλά θεωρούμε ότι είναι ανάγκη και νομίζω ότι το λέω εξ ονόματος όλων να απαντήσουμε στους ε, πολίτες οι οποίοι είναι αντικείμενο συμπεριφοράς ε, καθόλου σωστής. Υπάρχει απάντηση του Ισπανού Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος η οποία εστάλει πέρσι στην Επιτροπή μας ε, και εκεί αναφέρονται κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες ε, λογικά θα έπρεπε να ενταχθούν σε αυτή την πρόταση τροποποίησης που άκουσα να αναφέρεται σήμερα. Ίσως θα πρέπει να το αναφέρουμε. Υπάρχει και μία έκθεση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, η έκθεση Άουκεν, η οποία δυστυχώς δεν είχε τη συνέχεια που θα περιμέναμε και ε, θεωρούμε ότι το Κοινοβούλιο νομιμοποιείται να ζητήσει αναγνώριση ε, των δικαιωμάτων ε, τα οποία πρεσβεύει και υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά αναπάντητα ερωτηματικά. Ε, νομίζω ότι υπάρχει πολλή δουλειά για την Επιτροπή μας και τουλάχιστον μέσω των μέσων που διαθέτουμε κάτι θα μπορέσουμε να κάνουμε και θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με τους πολίτες που ζητούν την παρέμβαση του Κοινοβουλίου μέσω της Επιτροπής μας. Εάν συμφωνείτε λοιπόν για αυτό και για τα υπόλοιπα θέματα τα οποία ίσως δεν ανέφερα, θα ήθελα να σας ε, ζητήσω ε, να αποφασίσουμε αργότερα επί του θέματος. Απευθύνομαι στους συναδέλφους τώρα. Αναστέλλεται λοιπόν η απόφαση. Θεωρείται δεδομένο ότι οι αναφορές αυτές παραμένουν όλες ανοιχτές ε, και απόφαση θα ληφθεί στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών. Ευχαριστώ όλους τους παρεστημένους και ζητώ συγγνώμη για τυχόν παραλήψεις μου. Ο κύριος Γιάρ, επί της διαδικασίας, παρακαλώ. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να κάνω μια πρόταση. Επειδή είναι επίγον το θέμα. Αύριο το πρωί οι συντονιστές θα συναντηθούν και μπορούμε να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Αν έχουμε χρόνο βέβαια. Όχι. Δεν μπορείς. Τέλος εντάξει. Με το κανονικό χρονοδιάγραμμα λοιπόν θα συνεχίσουμε, αφού δεν μπορούμε να συναντηθούμε αύριο το πρωί. Την εκτιμώ την πρότασή σας, αλλά δυστυχώς ε, δεν γίνεται μάλλον. Θα δούμε κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα ε, για το μέλλον. Ευχαριστώ όλους τους παρισταμένους λοιπόν και να περάσουμε τι αναφορές που έχουμε στο επόμενο σημείο. Αναφορές οι οποίες παρουσιάστηκαν Συγγνώμη, η αναφορά μου λένε να περιμένουμε ένα-δυο λεπτά για να μπορέσουμε να έχουμε λίγο ησυχία για να αποχωρήσουν. Ε, διακοπή για δύο λεπτά. per Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μας να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, σας παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Λοιπόν, Σημείο 18. Δίνω απευθεία το λόγο στον πρώτο ε, αναφέροντα, το Λουκ Χιούμπνερ. Είναι παρόν? Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Bonjour, euh, voilà nous sommes... Euh, Καλημέρα. Είμαι εδώ εξ ονόματος μιας ένωσης, DCO No Merci. Πρόκειται για εκλεγμένους αντιπροσώπους, για ενώσεις, συλλόγους, όπως ε, Αλζάς Ματιό, προστασία του περιβάλλοντος στην Αλσασία. Είμαι ο Λουκ Ιμπέρ, αντιπρόεδρος της Αλζάς Νατιούρ και μέλος ε, του Συλλόγου No Merci. Είναι εδώ μαζί μου και ο Ντουάν Βέρτνερ. Θα δώσω το λόγο στο νομικό μας σύμβουλο, ο οποίος θα σας μιλήσει για τα τρία σημεία στα οποία παραβιάζεται η κοινοτική οδηγία. Ποιοι είναι οι στόχοι μας και γιατί είμαστε αντίθετοι με τον αυτοκινητόδρομο. Εδώ και 12 χρόνια, από το 99 δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει τη μάχη μας κατά αυτού του έργου. Όντως υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή του Στρασβούργου και θα πρέπει να βρεθούν λύσεις. Βλέπουμε όμως ότι η λύση που προτείνεται είναι ένα παλαιό σχέδιο αυτοκινητοδρόμου που υπάρχει από το 1970 και από τότε έχει ξεκινήσει μια μάλλον τεχνική συζήτηση για το πώς θα υλοποιηθεί το έργο αυτό. Σήμερα ο Σύλλογός μας δέχεται κάποιες ε, δύσκολες λύσεις. Βλέπουμε όμως σιγά σιγά ότι οι τεχνικές μελέτες δείχνουν τη μη βιωσιμότητα του έργου που προτείνουν οι αρχές. Εδώ και 12 χρόνια λοιπόν έχουμε αντιτεθεί και πριν δώσω το λόγο στο συνάδελφο που θα μας μιλήσει για τις νομικές πτυχές, θεωρώ ότι οι φάσει της λεγόμενης διαβούλευσης και μία εμπειρογνωμοσύνη ανεξάρτητη που έχει υποβληθεί δείχνει ότι οι υπηρεσίες του κράτους η νομαρχία μας βοήθησαν, μας στήριξαν, χρηματοδοτώντας αυτή την ανεξάρτητη μελέτη από την εταιρεία, τη γερμανική εταιρεία TICAR. Τα συμπεράσματα αυτής της έκθεσης είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Τα σημεία συμφόρησης περιγράφονται με το μαύρο χρώμα και μπορούμε να επιλύσουμε το θέμα χωρίς τον αυτοκινητόδρομο που προτείνουν οι αρχές. Η εμπειρογνωμοσύνη, η μελέτη της εταιρείας TTCAR μας έδειξε ότι υπάρχει τρόπος να επιληθούν τα προβλήματα γιατί το προτινόμενο έργο δεν ξεπερνάει τις δυσκολίες, δεν λύνονται δηλαδή τα συγκεκριμένα προβλήματα και θα συνεχίσει να υπάρχει συμφόρηση και μετά την κατασκευή του έργου. Αυτά όσον αφορά την ανεξάρτητη αυτή έρευνα που έγινε, τη μελέτη. Έγινε επίσης και μία δημόσια μελέτη. Εδώ και 10 χρόνια ακούμε όλες τις αρχές να μας λένε ότι πρέπει να γίνει αυτό το έργο, αυτός ο αυτοκινητόδρομος, γιατί θα λυθούν όλα τα κυκλοφοριακά προβλήματα του Στρασβούργου. Βλέπουμε ότι και οι γερμανικοί σύλλογοι μας στηρίζουν σήμερα. Η πόλη του Στρασβούργου ο Δήμος θεωρεί ότι πρόκειται για μία λανθασμένη λύση, μία εισφαλμένη λύση σε ένα υπάρχον πρόβλημα. Ακόμα λοιπόν και η αρχή που αρχικά πρότεινε, η Δημοτική Αρχή που πρότεινε αυτό το έργο, σήμερα είναι αντίθετη. Έχουμε ζητήσει από όλους τους πολιτικούς ε, της περιοχής μας να ταχθούν η Κατρίν Τρότμαν, οι σοσιαλιστές δηλαδή, είναι κατά, η πράσινοι επίσης και ο Γιώζεφ Ντόλ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, μας έγραψε αναφέροντας την αντίθεσή του στο πρόγραμμα αυτό. Θεωρούμε λοιπόν ότι και η μελέτη κόστος ωφέλειας όσον αφορά τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις που είναι σημαντικές θα μπορούσε να γίνει δεκτή εάν και εφόσον ε, επιλύονται τα θέματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, κάτι το οποίο σήμερα ξέρουμε ότι δεν θα γίνει. Δίνω μέσω στο λόγο και στο νομικό μας σύμβουλο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ματσόνη, καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Όπως είπε και ο Λούκα Ιμπνέργα, Μιλάμε εδώ πέρα για ένα αυτοκινητόδρομο μήκους 24 χιλιόμετρων που δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Μάλιστα υπάρχει και ένα διάταγμα το οποίο προβλέπει την κατασκευή του. Το θεωρούμε ότι βάλλονται καταρχάς εξή οδηγίες. Μία πρώτη οδηγία είναι αυτή που λέει ότι όταν από την κατασκευή ενός έργου πλήττεται ένα γειτονικό κράτος, τότε μπορεί, προβλέπεται, το γειτονικό αυτό κράτος να κάνει μία προσφυγή. Αναφέρομαι εδώ πέρα προφανώς στη Γερμανία και καταλαβαίνετε ότι το έργο αυτό θα επηρεάσει στην ουσία έμεσα και άμεσα τη χώρα αυτή όσον αφορά την κυκλοφοριακή συμφόρηση αλλά και τις επενδύσεις στη χώρα αυτή. Επίσης το σχέδιο αυτό για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου καταλήγει τελικά σε ένα δάσος στη Γερμανία και θα επηρεαστεί κατά αυτόν τον τρόπο και το περιβάλλον. Το ζήτημα αυτό έφτασε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας ακριβώς επειδή δεν έγινε σεβαστή αυτή η οδηγία και δεν ήταν επομένω το έργο αυτό έργο κοινή ωφελία. Στη συνέχεια βάλετε και η οδηγία εκείνη που να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος από την κατασκευή ενός έργου. Η Γαλλική Δημοκρατία δεν συνόδευσε την πρώτη κατασκευή του έργου αυτού κοινή οφειλίας από ένα σχέδιο περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έχουμε και επίσης την οδηγία 9243 όσον αφορά τον φυσικό οικότοπο, η οποία πλήττεται από την κατασκευή του έργου αυτού, καθώς επίσης και προστασία συγκεκριμένων ειδών όπως είναι ο κρικητός, καθώς επίσης και ο πράσινος φρύνος, ήδη τα οποία θα εκλείψουν από την κατασκευή αυτού του αυτοκινητοδρόμου. Βλέπουμε λοιπόν ότι πέρα από τις άμεσες αυτές επιπτώσεις υπάρχει και το ζήτημα της ε, μη χρησιμότητας κατασκευής ε, του έργου αυτού, καθώς επίσης και το έργο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως έργο κοινή ωφελίας όπως διατείνεται η Γαλλική Δημοκρατία. Απευθυνόμαστε λοιπόν εδώ πέρα στους ε, βουλευτές, εκπροσώπους των Ευρωπαίων πολιτών, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τις αρμοδιότητες που έχουν για να μην κατασκευαστεί το έργο αυτό, καθότι δεν παρουσιάζει κάποια χρησιμότητα ούτε κοινή ωφέλεια. Σας ευχαριστώ κύριε Ματσόνη, καθώς επίσης ευχαριστώ και τους βουλευτές για την προσοχή τους. Ε, ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Οι αναφέροντες συνόψησαν πολύ καλά την υπόθεση αυτή. Θα ήθελα και εγώ να δώσω κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά τα είδη στα οποία αναφερόμαστε και θα αναφερθώ λίγο περισσότερο από την όλη υπόθεση. Όσον αφορά λοιπόν την οδηγία για τους φυσικούς οικότοπους, αναφερόμαστε εδώ πέρα κυρίως στον κρικητό, ένα είδος όπου, που ευδοκιμεί κυρίως στην Αλσατία, παρουσιάζει πολύ σημαντική μείωση το είδος αυτό, μόλον ότι έχουν ληφθεί πάρα πολλά μέτρα προστασίας του. Οι απειλές για το είδος αυτό προέρχονται κυρίως από τις γεωργικές πρακτικές, καθώς επίσης και από τη γενικότερη τροποποίηση του φυσικού ενδιατήματό του. Έπειτα έχουμε και τον πράσινο φρύνο, που προστατεύεται και αυτός από την οδηγία για τους φυσικούς οικότοπους και πάλι το είδος αυτό εμφανίζεται κυρίως στην Αλσατία και θα επηρεαστεί πιστεύουμε την κατασκευή αυτού του αυτοκινητοδρόμου. Και εδώ πέρα το είδος αυτό απειλείται από τον κατακαιρματισμό του φυσικού κοτόπου του και από την τροποποίηση του περιβάλλοντος. Υπάρχει και το είδος Pelobat Brown, το οποίο βρίσκεται και αυτό κυρίως στην Αλσατία. Αναφερόμαστε λοιπόν εδώ πέρα σε τρία ζωικά είδη τα οποία απειλούνται. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στις ευρωπαϊκές διατάξεις που σχετίζονται με το με την υπόθεση αυτή. Ο κύριος Ιμπέρ ε, αναφέρθηκε σε τρεις οδηγίες οι οποίες φύγονται. Ε, Θα ξεκινήσω από την 42-2001 ε, και κυρίως από το άρθρο 7 της οδηγίας αυτής. Εδώ πέρα αναφερόμαστε στις, στα οδικά δίκτυα τα διασυνοριακά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει παραβίαση της οδηγίας αυτής που έχει ως στόχο να υποβάλλονται όλα αυτά τα προγράμματα για κατασκευή έργων τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν το περιβάλλον, να υποβάλλονται στην διαδικασία ανάλυσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε ένα σχέδιο και όχι σε ένα πρόγραμμα. Επομένως, ενδεχομένω να υπάρχει ένα πρόβλημα, ένα λάθος όσον αφορά τον εντοπισμό της οδηγίας αυτής. Η οδηγία 85337 που έχει να κάνει με τις ε, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή έργων, πάλι στο άρθρο 7 αναφέρεται στην διασυνοριακή διάσταση κάποιων έργων, όντως εδώ πέρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την οδηγία αυτή. Στην περίπτωση εκείνη που αναφέρον θα θέλει να χρησιμοποιήσει την ε, οδηγία αυτή και να κάνει αναφορά σε αυτή την οδηγία, μπορούμε να αναφερθούμε στα ακόλουθα σημεία. Πρώτον, ξεκίνησε μία διαδικασία καταγγελίας για το άρθρο 7, για παραβίαση του άρθρου 7, η οποία έγινε το 2010 και χρησιμοποιήθηκε το επιχείρημα ότι δεν είχαν συμβουλευτεί οι γαλλικές αρχές, τις γερμανικές αρχές. Βέβαια, δεν μπορούμε εμείς να εντοπίσουμε κάποια παραβίαση του άρθρου 7 της οδηγίας αυτής. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι το Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας το 2008 έλαβε μια προσφυγή για την ε, κατάργηση του, ε, της κατασκευής του έργου αυτού, της ε, διάταξης εκείνης της κρατικής η οποία προέβλεπε την κατασκευή του έργου αυτού. Το Μάρτιο όμως του 2010 το Συμβούλιο Επικρατείας απόφασή του είπε ότι στα πλαίσια της υπόθεσης αυτής και από τα επιδεικτικά στοιχεία δεν προκύπτει κάποια αρνητική επίπτωση όσον αφορά τις εικαζόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη Γερμανία. Όσον αφορά τώρα τις διασυνοριακές διαβουλεύσεις, η αναφορά δεν δίνει κάποια περαιτέρω στοιχεία που θα επέτρεπαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντοπίσει παραβίαση των κοινοτικών οδηγιών. Όσον αφορά τώρα την δεύτερη αυτή καταγγελία, τον δεύτερο ισχυρισμό που έχει να κάνει με το άρθρο 6 της οδηγίας όσον αφορά την αξιολόγηση των επιπτώσεων ορισμένων έργων στο περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι ε, η ε, υποβολή των αναλύσεων αυτών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αναλύθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας στη Γαλλία το 2008. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ωστόσο θα έρθει σε επαφή πάλι με τις γαλλικές αρχές προκειμένου να φανεί αν τελικά υπήρχε κάποια γαλλική αρμόδια αρχή επί του περιβάλλοντος η οποία γνωμοδότησε για την κατασκευή του έργου αυτού και τι επιπτώσει που θα μπορούσε το έργο αυτό να έχει στο περιβάλλον. Όσον αφορά την καταγγελία αυτή που έχει να κάνει με την κοινοτική οδηγία για το φυσικό οικότοπο και το άρθρο 12, στο άρθρο 12 προβλέπεται ότι τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να δημιουργήσουν ένα αυστηρό σύστημα προστασίας για τα ζωικά αυτά είδη τα οποία ε, ε, εμφανίζονται στο παράρτημα 4 της Οδηγίας. και απαγορεύεται κατά αυτόν τον τρόπο η καταστροφή, των ε, φυσικών οικότοπων ή των χώρων ανάπαυσης των ε, ε, ειδών αυτών. Ο κρικιτός λοιπόν, ο πράσινος φρύνος και το Pelobite μπράν, που είναι είδος και αυτό φρύνου, περιλαμβάνονται στο παράρτημα 4 της οδηγίας αυτής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε προσφυγή κατά της Γαλλίας ε, στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη σεβασμό του άρθρου 12 της ε, κοινοτικής οδηγίας για το φυσικό οικότοπο, κυρίως για το είδος κρικητός. Θα μπορούσε αυτό να ισχύσει και για τα άλλα είδη, δηλαδή τον πράσινο φρύνο και το άλλο είδος φρύνου. Στι 9 Ιουνίου θα έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει λοιπόν εκ νέου την αναφορά υπό το φω της δικαστικής απόφασης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα θα αναφερθώ στο θέμα αυτό γιατί νομίζω ότι οι αναφέροντες αλλά και η Επιτροπή παρουσίασαν με πολλές λεπτομέρειες την ε, υπόθεση αυτή. 15 μέρες μετά την ε, νέα στρατηγική για την βιοπικιλομορφία, βλέπουμε ότι η στρατηγική μας έχει αποτύχει. Εμείς, σαν μέλη του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου, έχουμε αποτύχει Καταλαβαίνετε από από τη μία μεριά έχει αποδειχτεί η αναποτελεσματικότητα, η αχρηστία ενός τέτοιου έργου και αυτό είναι, αν θέλετε, και συμβολικό για το πόσο έχουμε αποτύχει στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την βιοπικιλότητα. Πρέπει να το λάβουμε φοβερά πολύ σοβαρά υπόψη μας αυτό, διότι η φοβερή μας φιλοδοξία αυτή τη στιγμή έχει βρεθεί μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Σήμερα κινδυνεύουμε να βρεθούμε μπροστά στο φαινόμενο της εξαφάνισης αυτών των ειδών, αλλά και του ευρωπαϊκού μοντέλου αγροτικής ανάπτυξης, αυτό είναι κάτι που έχει ξεκινήσει ήδη από το 1970. Είναι λοιπόν αυτό συμβολικό γιατί πριν από 30 χρόνια το χάμστερ αυτό υπήρχε παντού. Σήμερα οι σύλλογοι προστασίας του περιβάλλοντος έστειναν παγίδες όταν ήταν μικρά παιδιά και πρόκειται για ένα θηλαστικό το οποίο καταφέραμε μέσα σε μία γενιά να το εξαφανίσουμε. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά να είμαστε όλοι πολύ απαιτητικοί, να δείξουμε συνοχή, να επιμείνουμε στις θέσεις μας, να ζητήσουμε από το γαλλικό κράτος να επιμείνει, να ανατρέψουμε την σημερινή τάση γιατί πραγματικά αυτά τα είδη απειλούνται και είναι σχεδόν, σχεδόν εξαφανισμένα και στη Γαλλία αλλά και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος άλλος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Ωραία. Να δώσουμε χρόνο απάντηση στον εκπρόσωπο της ε, ΣΥΖΙΟ. Δύο λόγια μόνο για να απαντήσω στην Επιτροπή. Η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αφορά δύο πτυχές που αφορούν ε, το μεγάλο χάμστερ. Πρόκειται για θέματα που αφορούν την αστική επέκταση. Η Τζούλιαν Κόκοτ, εισαγγελέα του δικαστηρίου, υπενθυμίζει ότι οι πτυχές αυτές δεν αφορούν την παρούσα υπόθεση. Δηλαδή, ό,τι έχει σχέση με τις μεταφορές είναι θέματα που παραμένουν ανοιχτά. Γι' αυτό και ζητάμε σήμερα από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μας στηρίξουν και σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας, την τελευταία παρέμβαση. Επίσης θέλω να σας πω ότι οι έρευνες αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί και είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ακόμα δεν έχει ληφθεί η τελική απόφαση. Εγώ θα ήθελα απλώς να πω ότι ειλικρινά μπορούμε να αφήσουμε αυτήν την αναφορά ακόμη ανοιχτή, περιμένοντας και τη γαλλική κυβέρνηση και την Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που μπορούμε να ζητήσουμε και μπορούμε να το πετύχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω κάποιον να αντιτίθεται. Μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε την πρόταση του κυρίας Μπελιέ, την οποία υποστηρίζει και ο κύριος Μποστινάρου. Η αναφορά παραμένει ανοιχτή και ευχαριστώ τους αναφέροντες, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεργασία. Έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν με τα σημεία της ημερήσιας διάταξης ε, για το σημείο Β αναφορές για τις οποίες ε, προτείνεται να περατωθούν. Έχουν ε, ζητηθεί κάποιες αναβολές σε κάποια σημεία, πιο συγκεκριμένα οι αναφορές 25, 26, 27, 30, 36 και 40 και αναφορές 03 ε, του 2005, 1078 του 2009 και 568 του 2007 έχουν διατυπωθεί τα αιτήματα αυτά και εγκρίνεται η μερίσια διάταξη για το σημείο ε, Β με τις τροποποίησεις που πρότειναν οι συνάδελφοι και τις αναφορές που σας ε, είπα. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Πέρασε συνεδρία. Ευχαριστώ.